Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf die unterbrochene Sitzung. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Αρχίζουμε την συνεδρίασή μας. Σήμερα έχουμε ψηφοφορία δύο εκθέσεων. Ξεκινάμε λοιπόν με την έκθεση της κυρίας Ιβάνοβα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ετήσια έκθεση του 2010. Η συγγήτρια δεν είναι εδώ σήμερα και κατόπιν τούτου δεν μπορεί να τοποθετηθεί. Κατόπιν τούτου μπορούμε να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσως ε, με την ψηφορία. αν συμφωνείτε βέβαια και εσείς. Ε, δεν βλέπω να υπάρχει αντίρρηση. Τροπολογία 1. Εδάφιο Β. Ποιος συμφωνεί παρακαλώ να σηκώσει το χέρι. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1, συμβιβαστική 1, υπέρ παρακαλώ, κατά, ε, δύο αποχές, ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 καταπίπτει, Πάμε στην C2, συμβιβαστική 2, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9, υπέρ, είναι προφορική η τροπολογία αυτή. από τον συνάδελφο Ντόιτς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μια προφορική τροπολογία και αναφέρει ότι ενθαρρύνει τις χώρες με καλή δημοσιονομική πειθαρχία ε, και περιοχές σύγκλησης. Αυτή είναι η προφορική τροπολογία. Αντιρρήσει, παρακαλώ για αυτή την προφορική τροπολογία. Δεν βλέπω. Έτσι μπορούμε να ψηφίσουμε για την τροπολογία υπαριθμών 9. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος, ε, δεν ψηφίσαμε για την τροπολογία υπαριθμών 11. Πάμε πίσω στην ε, τροπολογία υπαριθμών 11. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές. Νομίζω αυτό πρέπει να το ελέγξουμε. Την 15 παρακαλώ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, έκλεισε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπερθμών 16. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. Ε, επαναλαμβάνουμε για την 16. Υπέρ παρακαλώ, κατά, νομίζω είναι σαφές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ή 17 παρακαλώ, ε, καταπίπτει, ε, πάμε στη συμβαστική 5, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 καταπίπτει. Όχι, δεν καταπίπτει, γιατί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 31 υπέρ κατά αποχές. Ε, για μένα δεν είναι σαφές. Ας ελέγξουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την 31. Για την 31 ψηφίζουμε. Για την 31 παρακαλώ, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Κάτσε να βάλουμε αυτό. Το έκλεισε. Το έκλεισε. Ωραία, καλύτερα έτσι. μου υπενθύμησαν ότι μπορεί να ψηφίσει είτε ο κύριος Μπάρτον είτε ο κύριος Έρενχάουζερ. Ένας από τους δύο μπορείτε λιγάκι να το διευκρινίσετε παρακαλώ. Ο κύριος Έρενχάουζερ είναι το πλήρες μέλος, εκείνος μπορεί να ψηφίσει. Συνεχίζουμε λοιπόν με την τροπολογία 33 παρακαλώ, όχι έκανε λάθος ο πρόεδρος, 32 παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 33 τώρα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ η 36 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 41 παρακαλώ. Τροπολογία 41. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 11 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ για τη 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε. Ε, οριακό το αποτέλεσμα. Και έχουμε δύο ψήφους χωρίς κάρτα. Άρα εγκρίνεται. Η 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι, όχι, ε, απορρίπτεται, ελέγχουμε παρακαλώ για την 47. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται λοιπόν. Η 48 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 49 υπέρ κατά αποχές ασαφές είναι το αποτέλεσμα για τη 49 ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά έκλεισε η ψηφοφορία εγκρίνεται η 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 51 αποσύρθηκε για την 52 μισό λεπτό υπάρχει εδώ ε, προφορική τροπολογία του Γκέρ Μπενιάν. Είναι μια τεχνική φύσεως τροπολογία, δηλαδή να αντικαταστήσουμε τη λέξη στα αγγλικά subsidies με τη λέξη funding. Αντιρρήσεις παρακαλώ δεν υπάρχουν. Ψηφίζουμε λοιπόν, ψηφίζουμε ως τροποποιήθηκε η τροπολογία, η 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 55 παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 56 προφορική τροπολογία, καταπίτη, 58 υπέρ, κατά, κατά παρακαλώ, αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 14 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πάμε τώρα ε, στις γνωμοδοτήσεις. Της ε, ΔΕΒΕ, υπαρτμόν 1, Επιτροπή Ανάπτυξης, μπορούμε να ψηφίσουμε συνολικά για την 1-2-3 της ανάπτυξη υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Η τροπολογία 4 της Επιτροπής Ανάπτυξη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 5 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, ΔΕΒ6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, ΔΕΒ7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρινεται δβ ΔΕΒ8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε ε, συνολικά για την 9 μέχρι την 12 υπέρ αποχές ε, εγκρίνονται. Πάμε τώρα στην γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, της ΕΚΟΝ. ΕΚΟΝ 1 ναι. υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. ΕΚΟΝ 2 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. ΕΚΟΝ 3 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Εκον 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκον 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκον 6 υπέρ Μισό λεπτό έχει καταπέσει. Πάμε στην έκον 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται από την 7 ε, μέχρι την 11, 7 ε, μέχρι 11 μπορούμε να ψηφίσουμε για όλες αυτές, ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Έκον 12 και 13 καταπίπτουν, οι 14... Τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε συνολικά για τις Τροπολογίες 14 μέχρι 26. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Ε, της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, η NV3 μέχρι την 7 unblock υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. NV8 υπέρ κατά αποχές ασαφές το αποτέλεσμα. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ την NV8. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Ο Γιάνν ε, ψήφισε υπέρ. Εγκρίνεται. Ναι. NV9. Από την 9 μέχρι την 12 unblock ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τώρα, ψηφίζουμε για το σύνολο του ε, σχεδίου ψηφίσματος, ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έκλεισε η ψηφοφορία. Έτσι λοιπόν εγκρίνεται η έκθεση αυτή. Συγχαρητήρια στην κυρία Ιβάνοβα, την εισηγήτρια. και τώρα συνεχίζουμε Έκθεση Ριβελίνη. Ο εισηγητής, μήπως ε, θέλει να πει κάτι πριν να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα επιθυμούσα αλφή να αποδώσουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την πρόταση γιατί βρισκόμαστε ε, σε μια βαθιά κρίση και κάνω έκκληση σε όλους τους ευρωβουλευτές ε, διότι η κρίση δεν πλήττει στην Ευρώπη μόνο μία χώρα είναι μία κρίση που μαστίζει το σύνολο της Ευρώπης μία κρίση η οποία κατά κάποιον τρόπο επεκτείνεται και σε άλλες χώρες γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι τα μέτρα που αφορούν τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τα μέτρα αυτά ε, θα πρέπει να επεκταθούν σε όλες τις ε, χώρες της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν κρίση. Το να τα περιορίσουμε σε μία και μόνο χώρα, αυτό είναι άδικο. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνομαι στο αίσθημα δικαίου όλων των συναντέλφων. Πιστεύω ότι οι τροπολογίες από την 6 μέχρι την 9, όπως είπε και η Γραμματεία, είναι όλες οι ίδιες και γι' αυτό ε, μπορούμε να ψηφίσουμε unblock από την 6 μέχρι την 9. Ευχαριστούμε κύριε Ριβελίνη. Λέω ο πρόεδρος, ο κύριο Ριβελίνη, τροπολογίες 6 έω 9, να ψηφιστούν unblock. Συμφωνείτε ή μήπω επιθυμείτε ε, ξεχωριστή ψηφοφορία για κάθε μία από αυτε Αν ε, ψηφίζουμε unblock, ε, ξεκινάει ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για την 6 έω την 9, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, απορρίπτονται έλεγχος όμως ηλεκτρονικός 6 έως 9 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Έκλεισε ψηφοφορία. Ε, Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρία υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Παρακαλώ να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία αριθμός 3. Πέρας της προφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 13. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 παρακαλώ, υπέρ ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 13, θέλετε για τη 13, εντάξει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη 13. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Λάθος έκανα. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Η τέσσερα τώρα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεν εγκρίνεται. Επαναλαμβάνουμε για την 4. Υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Τώρα κατά. Όχι, είναι σαφές. Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ε, για την 4 ε, ψηφίζουμε. Για την 4 παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφορία. οριακό το αποτέλεσμα, αλλά πράγματι απορρίφθηκε. 13 με 12 είναι το αποτέλεσμα. Μερικές φορές είναι δύσκολο βέβαια να δει κανείς εδώ από την έδρα. Γι' αυτό και έχουμε τον ηλεκτρονικό έλεγχο ή 14. Υπέρ της 14 παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολογή 8. Υπέρ παρακαλώ. Κατά Άποχες. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Παρακαλώ, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία αριθμός 8. Ψηφίστε. Πέρας της Να Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Πάλι θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία αριθμό 10. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότηση με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ο εισηγητή όμω έχει κάτι να πει. Παρακαλώ κύριε Ριβελίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι η πρόταση του εισηγητή υπέρ της διεύρυνσης ε, της ισότητας της δικαιοσύνης στην Ευρώπη, αυτή δεν έγινε δεκτή. Βεβαίως ε, εγώ ευχαριστώ τους ε, συναντέλφους ε, και δέχομαι τις δημοκρατικές αποφάσεις, αλλά εγώ θα καταψηφίσω την έκθεσή μου γιατί η δυνατότητα να δοθεί αυτή, η ευκαιρία να δοθεί αυτή η δυνατότητα σε όλες τις χώρες είναι κατά του δικού μου του αισθήματο δικαιοσύνη. Εγώ λοιπόν θα καταψηφίσω τη δική μου την έκθεση. Mm. Βεβαίως δεχόμενος και σεβόμενος τα, τις δημοκρατικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε κύριε Ριβελίνη. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της, ε, του σχεδίου γνωμοδότησης. Μπορείτε να ψηφίσετε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα τη ψηφοφορίες. Δεν λειτουργήσε το μηχάνημα. Να το επαναλάβουμε τότε. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 14-10. 15? Όχι. 14-11 είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Καλώς. Ψηφίσαμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Congratulations. Συγχαρητήρια. Όχι στον εισηγητή, τι να πω, στην επιτροπή μας. Ναι. Δεν ξέρω. Dann geht es weiter auf Deutsch, aber in der Abstimmung Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα γερμανικά. Βέβαια, στην ψηφοφορία προτίμησα να μιλήσω αγγλικά. Nach einem kurzen Moment μετά από έτσι ένα μικρό διάλειμμα που κάναμε. Συνεχίζουμε τώρα με την ημερήσια διάταξη, με το σημείο υπερτιμών 11 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για το σημείο υπερτιμών 11 για τον Γενικό Προεπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισηγητής μας είναι ο συνάδελφος Μπόκουσλαβ Λιμπεράτσκι και θα ήθελα να του δώσω το λόγο. Παρακαλώ κύριε Λιμπεράτσικη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη ευχαρίστηση θα σας παρουσιάσω την απαλλαγή 10 Έχουμε λοιπόν την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Επίσης, ε, ακούσαμε και την τοποθέτηση διαφόρων. Ε, είδαμε και το ερωτηματολόγιο του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Βέλε. Πήραμε την απάντησή του και είχαμε και πάρα πολλές συζητήσεις. Επίσης, Συζητήσαμε και με την κυρία Ρουτ Μπέρεντ και με έναν από τους αντιπρόεδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ συναντήθηκα και με το Σκιώδη συγκητή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Η τελευταία συνάντησή μας έλαβε χώρα εχθές και ευχαριστώ πάρα πολύ ε, και όλους τους άλλους γιατί ε, ήρθατε πάρα πολύ στη συνάντηση αυτή. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι δύο θέματα ε, και στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ. κυρία Ιβάνοβα, η οποία δυστυχώς ε, ασθενεί, ε, είπε μερικά σημαντικά πράγματα και είπε τα εξής. Ε, αναφέρθηκε στο θέμα της κλοπής απογραφία, Αναφέρθηκε στην ασφάλεια του πάρκινγκ, του χώρου στάθμευσης και ε, επίσης και στους ε, δημοσιογράφους ε, που έρχονται για κάποιο λόγο στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ τον κύριο Ρόμπραντ, ευχαριστώ τους συνεργάτες μας και θα ήθελα και εγώ να θίξω δύο θέματα που ήδη ανέφερε ο κύριος Ρόμπραντ. Θα θίξω την ψηφιοποίηση του Κοινοβουλίου, της υπηρεσίας μετάφρασης και ένα τρίτο θέμα που το έθιξε ο κύριος Ντόμπραντ, δηλαδή το κατά πόσον οι εισηγητές μας ε, μπορούν ε, να αποκτούν ένα να εγγράφονται στη μερίσια διάταξη της Ολομέλειας ως ειδικό θέμα. Δεύτερο τώρα σημείο. Το Κοινοβούλιο ε, εργάζεται όλο και πιο αποτελεσματικά όσον αφορά στις υπηρεσίες του και ας μην ξεχνάμε ότι έχει τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία συνθήκη έχει επιφέρει πολύ σημαντικές αλλαγές. Οφείλουμε λοιπόν να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν τομείς όπου είναι απαραίτητο ε, να πράξουν βελτιώσεις όπως στις ε, αγορές, ε, στην ασφάλεια, στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους ευρωβουλευτές και στην πολιτική ακινήτων. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες Έχετε την έκθεση μπροστά σας και να δούμε τώρα τι θα μας πούν οι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος, και θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων, σε εκπροσώπους μάλλον, η κυρία Γκρέσλε. Εγώ μιλώ εξ ονόματος της ε, ασθενούς ε, κυρίας Ιβάνοβα, η οποία μου έδωσε ένα σημείωμα να το παρουσιάσω. Βεβαίως θέλουμε να ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Λιμπεράτσκι, τον νέο κοσμήτορα. Και επιτρέψτε μου και μία προσωπική παρατήρηση. Κύριε Λιμπεράτσκι, στη σύγκρουση συμφερόντων που θα εμπλακείτε ε, προφανώς γιατί τώρα ε, με την ιδιότητά σας ε, του τώρα αυτή η σύγκρουση συμφερόντων δεν θέλω να συνεχιστεί. Εμείς ε, ως Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών ενδιαφερόμετα για μια ε, καλή αξιολόγηση. Μας άρεσε πολύ η έκθεσή σας και ε, αυτή είναι η έκθεση κοινοβουλίου, του κοινοβουλίου, η μόνη έκθεση τα τελευταία 8 χρόνια που δεν με ξενέβρισε, που τη δέχομαι. Ούτε και το πιστεύω βέβαια, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον εισηγητή, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βέλε, το ελεγκτικό συνέδριο και τον ε, εσωτερικό ορκωτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα θέλαμε να θίξουμε ορισμένα θέματα. Ένα εξ αυτών τον έφερε ήδη ο εισηγητή. Πρόκειται για το θέμα της ασφάλειας, κυρίως ασφάλεια στα γραφεία. Γιατί παρουσιάστηκαν φαινόματα κλοπής. Ε, δηλαδή, ορισμένοι συνάδελφοι ε, στις διακοπές των Χριστουγέννων ε, έχασαν πράγματα από τα γραφεία τους. Παρουσιάστηκαν απώλειες και θα ήθελα να γνωρίζω τι θα κάνει η διοίκηση για το θέμα αυτό. Μετά, η διαχείριση των χώρων στάθμευσης. Εξακολουθούμε να έχουμε περιορισμένη παρακολούθηση με κάμερες στους χώρους στάθμευσης ε, και πολύ περιορισμένη ασφάλεια, άρα δηλαδή προκύπτονται ε, ζημιές ε, στο χώρο στάθμευσης. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μερικές μερικοί, μερικοί με συγχωρείτε, χρειάζονται να μάθουν να οδηγούν πώς παρκάρουν στο χώρο στάθμευσης. Στη Γερμανία λένε ότι είναι γυναίκες αυτές κυρίως, αλλά δεν είναι, σας το λέω για να το πιστέψετε. Κατόπιν πρέπει να τεθεί το ερώτημα, μάλλον Το θέμα του νερού, κατά πόσον και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μετά, το θέμα των, της ανάθεσης ε, δημόσιων συμβάσεων. Ε, θα το διαβάσω στα αγγλικά, γιατί η κυρία Ιβάνοβα μου το έδωσε στα αγγλικά, ότι πρέπει να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις στο θέμα της ε, ανάθεσης συμβάσεων, αλλά το θέμα είναι ο εκ των έλεγχος, δηλαδή πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τη βέλτιστη σχέση ανάμεσα σε ποιότητα και τιμή. Ένα θέμα που μας απασχολεί συχνά είναι το γραφείο ταξιδίων. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα παράγραφος, ε, κύριε Λιμπεράσκη, στην έκθεσή σας, όμως η παράγραφος αυτή δεν απαντά τα προβλήματα που έχουμε. Η κυρία Ιβάνοβα διαπίστωσε ότι ένα εισιτήριο το οποίο αγοράζει κανείς από το γραφείο ταξιδίων κοστίζει 1.400 ευρώ και ε, στο ίντερνετ μπορεί κανείς να διαβάζει το ίδιο εισιτήριο για την ίδια θέση για 200 ευρώ. Και εγώ Συζήτησα με το Γραφείο Ταξιδίων και διαπίστωσα ότι οι ίδιοι άνθρωποι ε, στο ίδιο αεροπλάνο, στην ίδια θέση, από το ίδιο Γραφείο Ταξιδίων ε, πληρώνουν διαφορετικά χρήματα. Και διαπίστωσα επίσης ότι στους ε, ευρωβουλευτές χρεώνονται πιο ακριβά εισιτήρια από ό,τι στους συνεργάτες του Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό προκύπτουν σημαντικές διαφορές. Ε, κυρίως όσον αφορά το κόστος ε, των ταξιδιών ε, των αντιπροσωπιών. Ας πούμε, η ΑΚΕ πήγανε στην Κινσάσα και εκεί τα ίδια τα μέλη είχαν δαπάνες για πάνω από 5.000 ευρώ ε, και οι συνεργάτες 3.000 ε, ευρώ, το προσωπικό δηλαδή 3.000 ευρώ. Αυτά είναι ε, ανεξήγητα πράγματα, άρα δηλαδή για τη δική μας την καλή φήμη πρέπει να δούμε πώς υπολογίζει το γραφείο ταξιδίων το κόστος των εισιτηρίων των ευρωβουλευτών φοβάμαι ότι σε αυτό το γραφείο ταξιδίων η βέλτιστη τιμή δεν παίζει κανένα ρόλο. πήγαμε στην IT 5.300 ευρώ business κόστασε το εισιτήριο μου. Μα τι είναι αυτό, δεν τολμάει κανείς πια να ταξιδέψει. Ε, και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι προς όφελός μας ε, να ζητήσουμε καλύτερες τιμές από το Γραφείο Ταξιδίων. Μετά, ε, οι βοηθοί ε, που ταξιδεύουν και αυτοί στην Κινσάσα είχαμε 46 συνεργάτες και 25 βοηθούς αυτό κόστισε πάνω από 40.000 ευρώ. Αυτοί οι 25 βοηθοί κόστησαν πάνω από 40.000 ευρώ και αυτά τα πληρώνει ο φορολογούμενο. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για κοινοβουλευτική συνέλευση, αυτό αφορά κυρίω βουλευτέ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ταξιδεύουν και βοηθοί. Ε, φοβάμαι ότι πρέπει να το δούμε λιγάκι το θέμα αυτό. Ε, να δούμε τι ε, χρεώνουμε στο φορολογούμενο. Μετά το κτίριο Κόνατ Αντενάου στο Λουξεμβούργο. Στην, στο σχέδιο τη έκθεσή σα δεν γίνεται λόγο για την αύξηση των δαπανών. Για μας είναι σημαντικό να μας το εξηγήσετε αυτό. Ποιος αποφάσισε τι και τι δεν ισχύει πλέον. Ε, και εδώ νομίζω ότι πρέπει να το δούμε το θέμα. Και εγώ προσωπικά ενδιαφέρομαι να ενημερωθώ για τους νέους κανόνες για τις επισκέψεις των ομάδων. Ε, αλλάξαμε τους κανόνες, μειώνουμε το μέγεθος των ομάδων και έχω τώρα την εντύπωση ότι έχουμε περισσότερες ομάδες αλλά λιγότερους επισκέπτες. Άρα δεν κερδίσαμε τίποτα. Ε, με την ε, ίδια κούραση έρχονται λιγότεροι στο κοινοβούλιο από ό,τι παλαιότερα. Άρα δηλαδή και εδώ ε, θα σας ήμουν ευγνώμων αν εξετάζατε τους ισχύοντες κανόνες και το ποια είναι η αποτελεσματικότητά τους. Κατόπιν, έχουμε ένα πρόβλημα με την δομή ηλικιών. Ορισμένες, ορισμένοι συνεργάτες έχουν μέσο όρο πάνω από 50. Από τη Λιτουανία, τη Μάλτα, αυτοί έχουν μέσο όρο 35. Είναι λοιπόν φυσιολογικό να υπάρχει κάποια αύξηση προς τα πάνω στο όρο αλλά το θέμα είναι ε, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί νομίζω ότι δημιουργείται στους συνεργάτες μας δημογραφικό πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν θα σας ήμασταν ευγνώμονες να μας δώσετε εξηγήσει. Εμείς ε, θα καταθέσουμε κάποιες ε, τροπολογίες και κύριε Λιμπεράτσκι, ελπίζω αυτή τη φορά η έκθεση του Κοινοβουλίου να κυλήσει ειρηνικά. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας. Ευχαριστούμε κυρία Γκρέσλε, πάρα πολύ ζήτησαν το λόγο. Επτά νομίζω. Θα τους πάρω με τη σειρά. Ε, you, Ευχαριστώ πρόεδρε. Σε αυτή την εποχή της λιτότητας ζητούνται πάντοτε περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και εξοικονομήσεις. Δυστυχώς όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθυστερεί. Για το θέμα του αριθμού των υπαλλήλων Πρέπει να καταλάβουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχει αυξηθεί το κόστος λειτουργίας του, αυτό ήταν αναμενόμενο, αλλά οι αυξήσεις που προβλέπονται δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικότητες. Από την τελευταία διεύρυνση ο αριθμός βουλευτών έχει παραμείνει ο ίδιος σχεδόν, ενώ ο αριθμός των υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 58% τελείως δυσανάλογα ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη τον ε, μεγάλο αριθμό γλωσσών. Αν η Κομισιόν μειώσει το προσωπικό της, τότε το Κοινοβούλιο τι θα κάνει. Και έρχομαι τώρα στο επόμενο θέμα. Αν υπήρχαν λιγότεροι υπάλληλοι, λιγότερα κτίρια θα χρειαζόμασταν. Το Κοινοβούλιο αγοράζει ή δανείζεται 63 κτίρια, δηλαδή πάνω από το διπλάσιο του αριθμού τους προηγουμένως το 2002 και όλα αυτά πρέπει να θερμαίνονται, να προστατεύονται κτλ. Εδώ είναι ένα τομέα όπου μπορούν όντω να γίνουν εξοικονομήσει. Άλλο πρόβλημα είναι το δημόσιο χρήμα που δαπανάται για την αυτοπροώθηση της Ένωσης που μερικοί τη λένε προπαγάνδα. Ότι υπάρχει δηλαδή ένας ευρωπαϊκός λαός, δήμος. Και το Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο μέσω της Γενικής του Διεύθυνσης Επικοινωνίας όπως με το Europarl TV και άλλα σχέδια και προγράμματα και πρέπει αυτά να τα ελέγξουμε αυστηρότερα. Πάνω από 30 εκατομμύρια έχουν επενδυθεί από, για το web channel από το 2008 και μετά και ο ίδιος ο εισηγητής λέει ότι είναι πολύ λίγοι οι χρήστες ενώ πολύ ψηλό το κόστος. Εδώ που, εκεί που διαφωνώ είναι ότι Αντί να ζητούμε μείωση κατά 40% 8 εκατομμύρια το χρόνο του προϋπολογισμού του Web TV, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχει αποτύχει το πρόγραμμα αυτό και πρέπει να καταργηθεί. Τέλος, ο οίκος ευρωπαϊκής ιστορίας που ακόμα συζητιέται, δεν μας λένε για αυτό το θέμα ποιο είναι το συνολικό κόστος. 31 εκατομμύρια είχαν υπολογιστεί για να ανανεωθεί, να κενιστεί το κτίριο και άλλα ποσά 3 εκατομμύρια για εκθέσεις και λοιπά μέχρι το 2014. αλλά ερωτώ αυτό το κόστος ε, πώς εφαρμόζεται αυτές οι προβλέψεις γιατί υπάρχει κάτω από αυτό το κτίριο ο ποταμός Μάλμπεϊκ που είναι υπόγειος και μπορεί να του καταστρέψει τα θεμέλια. Χρειάζεται μια ακριβέστερη εξέταση και θέλω να προτείνω στον εισηγητή να καλέσουμε τον κύριο Πέτερινγκ που είναι υπεύθυνο του προγράμματος να έρθει στην Επιτροπή μας και να εξηγήσει ποιο είναι το ακριβές κόστος. Ευχαριστούμε ο κύριος Χάρτουγκ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για το έργο που έχει επιτελεστεί από το Ελεκτικό Συνέδριο και από τον εισηγητή. Χτες ήμουν στο Λουξεμβούργο και είχα την ευκαιρία να μιλήσω για την έκθεση αυτή με το Ελεκτικό Συνέδριο και αυτό που μου φαίνεται πολύ περίεργο είναι ότι υπάρχουν ε, ε, πολλά στοιχεία τα οποία δεν φαίνεται να είναι κανονικά που καταγράφονται. Ιδιαίτερα όμως με απασχολεί το τι θα κάνουμε με αυτή την έλλειψη κανονικότητας και στο κάτω-κάτω αυτή είναι η δουλειά μας. Εμείς είμαστε πολιτικοί και πρέπει να βασιστούμε στη δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου και να αποφασίσουμε κατά πόσο τα διάφορα σχέδια είναι αποτελεσματικά ή χρήσιμα ακόμα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι έφτασε η στιγμή η Επιτροπή Προϋπολογισμών να καθίσει και να κάνει αυτοκριτική και να δει όλα αυτά τα οποία έχει εγκρίνει. Ήτανε όντως σωστά ή μήπω όχι και πρέπει κάτι να σταματήσει. Τώρα, τι γίνεται στην Επιτροπή και στους επιτρέπους. Εκεί δεν κατάφερα να βρω ποιος είναι υπεύθυνο για διάφορα στοιχεία στον προπολογισμό. Θα ήθελα να το προσπαθήσουν αυτό και οι συνάδελφοι και να αλλάξει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. πρέπει να πούμε ε, στο συνάδελφο Χαρτούγκ ε, ότι η Επιτροπή, η Επίτροπη δεν υπέσαν καμία περικοπή στον προϋπολογισμό ε, και επιμένω σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό που είπατε, αλλά περιμένουμε λίγο για να μεταφραστεί, να ακουστεί σε όλους. Επόμενος, ο συνάδελφος κύριος Γκεμπράντι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή Λιμπεράσκη για τη δουλειά του. Νομίζω ότι είναι σημαντικό εδώ να μην κοιτάμε μόνο τι έγινε το 2010, αλλά να κοιτάξουμε λίγο τι συστάσεις κάναμε και παλιότερα, μετά το 2009, με τον κύριο Ήταλα για παράδειγμα, και να προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποια μαθήματα από το παρελθόν και να τα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Διάφορα θέματα θα μπορούσα να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα κάτι γενικό που αναφέρει και ο κύριος Λιμπεράτσκι. Είναι ότι βεβαίως και να γίνεται ξεχωριστή συζήτηση από την Ολομέλεια για την δικιά μας απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή, βεβαίως και για τον προπολογισμό δηλαδή της επόμενες χρονιάς, αλλά και για την απαλλαγή της προηγούμενης κάθε φορά γιατί νομίζω ότι πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη πολιτική σημασία στην απαλλαγή αυτή. Πρέπει τη συζήτηση να την κάνουμε πιο πολιτική από ό,τι είναι ε, προς το παρόν. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ε, αναλάβει την ευθύνη, να την αναθέσει δηλαδή στο σώμα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ολόκληρο. Δεύτερον, Πολύ θα ήθελα το Ελεκτικό συνέδριο να ετοιμάσει κάποια φορά μια ειδική έκθεση, ειδικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορούμε να το ζητήσουμε φυσικά, ε, αν δεν το αποφασίζει από μόνο του το Ελεκτικό συνέδριο. Και κάτι ακόμα. Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο βέβαια θα κοιτάξω να προσθέσω μέσω κάποιας τροπολογίας που θα υποβάλω. Πρόκειται για την ψηφιοποίηση των γράφων Νομίζω ότι υπάρχει κάτι πειραματικό που ήδη έχει ξεκινήσει με το σχέδιο e-Committee, ηλεκτρονική επιτροπή. Έτσι μειώνεται ε, το χαρτί, δεν τυπώνουμε πια τόσα πολλά χαρτιά και ηλεκτρονικά έχουμε τα έγγραφα. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι κάθε χρόνο επανέρχεται το θέμα της πληρωμής για τις ομάδες επισκεπτών. Πάντα ε, με ρευστό πληρώνονται οι επισκέπτες. Αυτό είναι το σύστημα των πληρωμών και νομίζω ότι δίνει μια στραβή εικόνα στο κόσμο το σύστημα αυτό πληρωμών που γίνεται στις ομάδες επισκεπτών. Τέλος, μια άλλη σύσταση που κάναμε πέρυσι και θα ήθελα να την ξανακάνουμε, είναι και για μας και για τους ευρωβουλευτές ε, δηλαδή, να μπαίνουμε κι εμείς στην είσοδο με ένα πάσο. Δεν βλέπω γιατί εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Το είχαμε αποφασίσει κάποια στιγμή. Φαίνεται να εξακολουθεί να είναι περίπλοκο. Θα έπρεπε και το Προεδρείο και οι κοσμήτορες να το αποφασίσουν, να υπάρχει αυτός ο κανόνας και καλό θα ήταν να το συμπεριλάβουμε αυτή τη φορά στην έκθεσή μας αυτή. Ευχαριστώ κύριε Φρουτσέσκοβα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Και πάνω απ' όλα θέλω να του πω ότι στην έκθεση αυτή εντοπίζονται διάφορα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους δικούς μας πόρους. Εγώ θα αναφέρω κάποια μόνο σημεία που πιστεύω ότι είναι σημαντικά στην έκθεση αυτή. Ήδη από πέρυσι μιλήσαμε για την έγκριση ε, στη διαχείριση του 2009 γι' αυτό. Πρόκειται για τις τιμές... Συγγνώμη, πρόκειται για τα βραβεία που δίνει το Κοινοβούλιο. Διορθώνω, μιλείτε, για τα βραβεία, όπως για παράδειγμα το βραβείο Λουξ. Εγώ πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει λόγο, δεν πρέπει να αξιολογεί τη δημιουργία, την κινηματογραφική ε, της ταινία. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κάτι διαφορετικό ή εν πάση περιπτώσει όχι για τα βραβεία πάντως. Γιατί εδώ διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια αύξηση 50% τελικά ε, στα βραβεία. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει σε τίποτα δεν προσθέτει τίποτα ούτε στην εικόνα του Κοινοβουλίου, ούτε βέβαια και στον Ευρωπαίο Φορολογούμενο που πρέπει να το πληρώσει. Το ίδιο ισχύει και για τα βραβεία που δίνουμε στους δημοσιογράφους. Θέλω τώρα να αναφερθώ λιγάκι στην τηλεόραση μέσω διαδικτύου που κοστίζει 1 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ποσό ιδιαίτερα υψηλό, πιστεύω. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ε, θεατών, δίνει υπερβολικά πολλά χρήματα για να γίνεται η αναμετάδοση αυτή των συνεδριασεών του. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε έναν άλλο τρόπο, κάτι που να παρακολουθούν πιο πολλοί άνθρωποι. Θα έπρεπε να απορρίψουμε την δαπάνη τέτοιων κονδυλίων που είναι για να βελτιωθεί η εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόνο, όπως είναι ο οίκος ιστορίας ή το μου. Τα ξέρουμε αυτά εδώ στην Επιτροπή μας. Αυτά είχα να πω. Κατά τα άλλα, α ναι, για την ασφάλεια ήθελα να προσθέσω κάτι. Η ασφάλεια στο πάρκινγκ. Ιδιαίτερα στο Στρασβούργο. Εκεί πραγματικά θα έπρεπε να ζητήσουμε να βελτιωθεί και οι υπηρεσίες που ασχολούνται με το πάρκινγκ στο Στρασβούργο πρέπει να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Για άλλη μια φορά, κάθε, με κάθε σεβασμό στο Στρασβούργο και στο κτίριό μας εκεί, πρέπει να πω ότι φέτος και εδώ θέλω να μιλήσω για τις υπηρεσίες που εξυπηρετούν εμά, του ευρωβουλευτέ. Τέσσερι μέρε το μήνα τι περνάμε εκεί στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό να το ξέρουμε ότι είμαστε εκεί από νωρί το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Λοιπόν, πώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα έχουμε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια της δουλειάς μας, της ολομέλειας που γίνεται εκεί, πώς θα μπορούσαμε να τρώμε καλύτερα, να έχουμε μεγαλύτερη επιλογή στις υπηρεσίες που παρέχουν διατροφή την εβδομάδα εκείνη. Δεν ξέρω. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε, να δημιουργήσουμε κάποιο είδους επιχείρηση για να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί ειλικρινά για τους ευρωβουλευτές και τους συνεργάτες μας δεν νομίζω ότι υπάρχει αρκετή επιλογή όσον αφορά το φαγητό στο Στρασβούργο, αλλά και γενικότερα σε εγκαταστάσεις που έχουμε στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ πολύ και για άλλη μια φορά θέλω να σας πω ότι στην έκθεση αυτή υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που και μένα με απασχολούν πολύ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λιμπεράσκη για την τόσο ενδιαφέρουσα έκθεσή του. Είναι γεμάτη ενδιαφέροντα στοιχεία και προτάσεις για το Μάιλον. Φαίνεται ότι υπάρχει μια βελτίωση. Για το θέμα της ασφάλειας πρώτα απ' όλα τώρα. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Στις παραγράφους 31 και 32 μιλάμε για ένα διαχειριστή κινδύνου. Αυτός ο διαχειριστής ε, κινδύνου είναι για την ασφάλεια φαντάζομαι. Είναι αυτός που διαχειρίζεται οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για την ασφάλειά μας. Έτσι δεν είναι. Αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λιμπεράσκη. Επίσης, δεδομένου ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα ασφάλειας, παρόλα αυτά έχει μειωθεί ο προπολογισμό που πάει στην ασφάλεια. Δεν υπάρχει μια αντίφαση. Θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε αυτό, πώς γίνεται. Άμα μειωθεί ο προπολογισμό, δεν θα υπάρχουν προβλήματα διαχείριση ε, του κινδύνου. Πώ θα το διαχειρίσουμε ακόμα καλύτερα τον κίνδυνο, πώ θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, διάφορα άλλα πράγματα τα έχουν ήδη ρωτήσει οι συνάδελφοι. Το επόμενο που θέλω εγώ να πω είναι αυτό που μιλάμε για ένα γραφείο σύνδεση που θέλουμε να έχουμε στην Ουάσιγκτον. Ωραία, μπορεί να είναι ε, ενδιαφέρον στις άλλες, στα άλλα γραφεία, τα εξωτερικά, το κοινοβούλιο μας πώς είναι παρόν, έχουμε στοιχεία, πόσο δηλαδή καλύπτεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα γραφεία αυτά τα εξωτερικά που έχουμε, όχι επιτροπή αλλά το κοινοβούλιο. Επίσης, μιλάμε και για ε, πρόσληψη υπαλλήλων από ορισμένε υπηκότητε. Μιλάμε για ένα δημογραφικό βάρο. Εγώ θέλω να έχω συγκεκριμένα, όχι τα ποσοστά, αλλά γιατί. Στην παράγραφο 54. Ποιο είναι ο λόγο για τον οποίο στο Κοινοβούλιο δεν έχουμε υπαλλήλου από αυτές τι χώρες τι οποίε αναφέρεστε. Υπάρχει κάποιος λόγος ή μήπω οι θέσεις που έχουμε να τους προσφέρουμε δεν τους ε, ενδιαφέρουν γιατί έχουν καλύτερη δημόσια υπηρεσία στις δικές τους χώρες και γι' αυτό δεν έρχονται εδώ. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους δεν έχουμε εδώ υποψηφίους από αυτές τις τέσσερις χώρες τις οποίες αναφέρετε εδώ. Κατά τα άλλα η εκθεσή σας μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη. Συγχαρητήρια και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γιάλα Σέντερ. Ο κύριος Απατσίτης παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα πράγματι. Έχει πολλές πληροφορίες. Αλλά ομολογώ ότι χαίρομαι που δεν ήμουν εγώ υπεύθυνο για την ανάλυση της δαπάνησης των της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι η Ευρώπη <clears throat> και ο κόσμος ολόκληρος ζουν μία σοβαρή κρίση και οι αρχές που είχαμε εγκρίνει προηγουμένως δεν μπορούν να διατηρηθούν όσοι είχαν Ίσως επαναλαμβάνω πράγματα που είπαν και άλλοι, αλλά μου φαίνεται αναπόφευκτο να γίνουν αλλαγές. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν πληρώνουμε μόνοι μας τα ναύλα μας, αλλά παρόλα αυτά συμφωνώ με την κυρία Γκρέσλερ, δηλαδή Νομίζω ότι το θέμα αυτό των αεροπορικών εισιτηρίων αφορά εκατομμύρια ευρώ που δεν χρησιμοποιούνται με τον καταλληλότερο τρόπο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά τα αεροπορικά του εισιτήρια. Έτσι κάνουν και οι ιδιωτικές εταιρείες πρέπει να έχουμε πάντοτε τα φτηνότερα δυνατά εισιτήρια για να μειώσουμε το κόστος. Άλλο πρόβλημα. Το γκαράζ, τα πάρκινγκ. Έχουν ληφθεί αρκετά παράλογες αποφάσεις και μπορούν εδώ τα πράγματα να βελτιωθούν σημαντικά. Σημαντικά. Παραδείγματο χάρη για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα και εδώ η κατάσταση δεν είναι καλή. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι τιμές της αγοράς και να βελτιώσουμε τα πράγματα. Έχουμε τρεις τόπους εργασίας, έτσι αποφασίστηκε κάποτε. να υπάρχουν τρεις τόποι εργασίας, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο. Πρέπει όμως κάποτε νομίζω να απαντήσουμε κάποτε στο ερώτημα γιατί ταξιδεύουν τόσα μέλη του προσωπικού μεταξύ των τριών τόπων εργασίας ενώ θα μπορούσαν όλα να γίνονται σε έναν. Έπειτα. Άλλο θέμα που με ανησυχεί και που πρέπει να το ξαναδούμε λεπτομερέστερα είναι το θέμα του, ταμείου εθελοντικής συνταξιο... του Εθελοντικού Ταμείου Συνταξιοδότησης που έχει έλλειμμα. <coughs> και αυτό με ανησυχεί. Και πρέπει να δούμε γιατί υπάρχει αυτό το έλλειμμα. Ο κύριος Σόνικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Λιμπεράτσικη για την έκθεσή του, αλλά να κάνω και μερικά σχόλια. Το βραβείο Λουξ του 2011 έχει και αυτό αυξήσει το κόστος λειτουργίας του. Από 300.000 ευρώ στα 375. το βραβείο αυτό το απονέμει, το δίνει το κοινοβούλιο. Είναι προφανώς κάτι χρήσιμο, αλλά είδα τα έργα που βραβεύονται. Ζήτησα μάλιστα να προβληθούν και στην Κρακοβία και δεν μπόρεσα δυστυχώς να το πετύχω. Δεν μπόρεσα να πετύχω τη μετάφρασή τους, τον υποτιτλισμό τους. Αν δαπανούμε τέτοια ποσά για να μην μπορεί καν μετά το έργο να μεταφραστεί, <coughs> τότε νομίζω ότι αποτυγχάνουμε. Η έκθεση αυτή είναι μια απαρίθμηση ευχών αλλά και επικρίσεων. Ζήτησα από τη διοίκηση το 25% της τιμής του βραβείου να χρησιμοποιηθεί και για τη δημιουργία ενός αρχείου του Κοινοβουλίου για την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα ακόμη να συνομιλήσω με τη Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας γιατί βρίσκω ότι είναι κάπως αλαζονική η στάση της. Το λέω ρητά, αλαζονική. Έπειτα και για τις κλοπές πρέπει κάτι να κάνουμε για τα Γιατί βρίσκω ότι και στο δικό μου γραφείο εκλάπησαν πολλά αντικείμενα και δεν μπόρεσα καν, καν λέγω, να επαληθεύσω αν ξαναβρέθηκαν αυτά τα αντικείμενα ή είναι στο γραφείο απολεσθέντων. Δεν μπόρεσα να το μάθω. Μπόρεσα Όσο για τα γραφεία πληροφόρησης που έχουμε, εκείνο της Βαρσοβίας ομολογεί ότι δεν γνωρίζει αν λειτουργεί αποτελεσματικά γιατί και οι ίδιοι ευρωβουλευτές οι Πολωνοί δεν μπορούν πάντα να έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση από εκεί. Πολλές φορές τα ναύλα μας αλλάζουν ξαφνικά. Είναι βέβαια και μεγάλος ο αριθμός των εισιτηρίων που πρέπει να εκδίδει το ταξιδιωτικό μας γραφείο και δεν μπορεί πάντοτε να εγγυάται την καλύτερη τιμή. Μπορεί. Δεν ξέρω μήπως το σύστημα θα ήταν να πληρώνει ο καθένας μόνος του και μετά να τον αποζημιώνουν ίσως να ήταν πιο αποτελεσματικές οι εξοικονομήσεις. Εγώ είμαι καινούριο στην Επιτροπή αυτή και δεν ξέρω ποια είναι τα ήθη, αλλά... αλλά να. Είχα διαβάσει, παραδείγματο χάρη, ότι σήμερα θα ψηφίζαμε στις 9.30 και μετά μου είπαν όταν ήρθα ότι είχε ήδη γίνει η ψηφοφορία. Θέλω να σεβόμαστε τα προγράμματα. Κοιτάξτε, όσον αφορά την ψηφορία, 9 η ώρα προβλεπόταν στην ημερησία διάταξη. Και μάλιστα αργήσαμε λιγάκι και κατά 10 λεπτά. Δεν ξέρω. Δηλαδή, στην ημερήσια διάταξη που σας ε, είχε σταλεί προβλεπόταν 9 η ώρα. Αλλά δεν ξέρω, αυτό μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε και με τη γραμματεία. Äh, Από ό,τι φαίνεται έχει γίνει κάποιο λάθος ε, στη γραπτή μετάφραση του κειμένου. Αυτό ε, πρέπει να το προσέξουμε, γιατί προφανώς ε, δεν μπορούν να έρθουν μέλη να ψηφίσουν. Εν πάση εγώ με την μερίσια διέταξη να έχω στα γερμανικά και εκεί αναφέρεται σωστά η ώρα. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, ε, έχουν ζητήσει πολύ το λόγο. Επτά. Θέλω μόνο να σας υπενθυμίσω ότι βεβαίως το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει το δικό του το προπολογισμό είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να εμφανιζόμαστε και ως πρότυπο. Πρέπει δηλαδή τα του οίκου να τα εξετάζουμε εξίσου αυστηρά όπως και άλλων οργανισμών. Γι' αυτό θεωρώ ότι η συζήτηση είναι πολύ σημαντική και ε, πρέπει να δώσουμε χρόνο στην εξέταση αυτού του θέματος. Όσον αφορά στην αποτελεσματική χρήση κονδυλίων, εδώ ε, πρόκειται ε, για τους στόχους μας που έχουμε θέσει, αλλά να τους επιτύχουμε με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ε, το θέμα των ε, ταξιδιών, των αποστολών, αυτό είναι θέμα αποτελεσματικότητας. αν πρέπει να πάμε επιτόπου πράγματι πρέπει να ταξιδεύουμε οικονομικά. Αυτό είναι ένα θέμα που ετέθη και πιστεύω ότι την αποτελεσματικότητα πρέπει πράγματι να την εξετάσουμε και θα ήθελα να παρακαλέσω συναδέλφου να έχουν κατά νου ότι έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά θέματα στην ημερησία διάταξη. Ο συνάδελφος κύριος Γκάια έχει ζητήσει το λόγο, μετά Ματιό Οντί και πολλοί άλλοι. Ο κύριος Γκάια έχει το λόγο καταρχήν. Ε, εγώ έλαβα σοβαρά αυτό που είπατε κύριε Πρόεδρε περί του περιορισμένου χρόνου και αποσύρω την παρέμβασή μου. Κυρία Ματιού. Θα είμαι τότε πολύ σύντομη, Πρόεδρε, αφού είναι έτσι. Μια που και ο κύριος Γκάγια παρετήθηκε. Θα αναφερθώ σε ένα μόνο σημείο. Πρώτα απ' όλα βέβαια θέλω να συγχαρώ για την εξαίρετη εργασία του τον εισηγητή και θέλω να επανέλθω στο θέμα των επισκεπτών. Βέβαια δεν ευθύνεται ο εισηγητής, αλλά εγώ θέλω να επανέλθω σε αυτό γιατί έγινε μεν μια μικρή προσπάθεια από πλευράς του Κοινοβουλίου, αλλά δεν είναι αρκετή. Οι ομάδες επισκεπτών, που βέβαια είναι πολύ σημαντικές, επισκέπτες δηλαδή και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολόκληρο, αλλά και για μας τους Ευρωβουλευτές, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να τους δείξουμε τι κάνουμε, να τους δείξουμε τη δουλειά μας, γιατί το Κοινοβούλιο είναι μια βιτρίνα για όλους τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Είναι σημαντικό η εικόνα που δίνουμε προς τα έξω. Όταν λοιπόν ένας υπάλληλο φέρνει τον ε, υπεύθυνο της ομάδας επισκεπτών για να πληρώσει και του δίνει σε ρευστό ένα πολύ σημαντικό ποσό που μπορεί να είναι 6, 7 μέχρι και 10 σε χαρτονομίσματα, νομίζω ότι δεν είναι καλό. Βγαίνει από εδώ κάποιος με ένα φάκελο, με ένα σωρό λεφτά μέσα Ειλικρινά, εγώ πιστεύω ότι η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή. Ορισμένοι υπεύθυνοι τέτοιων ομάδων επιχειρητών μου λένε Αχ, τι ωραία που περνάτε εσεί εδώ στι Βρυξέλλε, φεύγει με τα λεφτά στην τσέπη του. Ε, δεν είναι καθόλου καλή εικόνα αυτή που δίνουμε. Μερικέ φορέ πρόκειται για ομάδε επισκεπτών που έρχονται από πολύ χαμηλά στρώματα εισοδηματικά. Τα ποσά αυτά για αυτού είναι τεράστια. Δίνουμε πολύ άσχημη εικόνα. Λοιπόν, τι θέλω, θέλω το κοινοβούλιο όταν καλεί κάποιους επισκέπτες να μην δίνει ρευστό, αλλά να ε, αποζημιώνει για τα αεροπλάνα ή για τα λεωφορεία ανάλογα με το τι έρχονται και να πληρώνει από μόνο του τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια που έχει να πληρώσει. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι πιο περίπλοκο για το κοινοβούλιο ίσως, αλλά τουλάχιστον δεν δίνουμε αυτή την άσχημη εντύπωση που δίνουμε τώρα πιστεύω ότι είναι αντιπαραγωγικό και για τους ευρωβουλευτές αλλά και για το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε κάνει αρκετή προσπάθεια σε αυτό. Δεν έχει αλλάξει η εικόνα μας. Αυτά ήθελα να πω, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κυρία Ματιέ. Επόμενος, ο κύριος Οντί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα αναφερθώ στις πολιτικές δραστηριότητες των ε, υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι βέβαια δικαίωμα του κάθε πολίτη να έχει πολιτικές δραστηριότητες στις χώρες του. Όμως, πώς ελέγχουμε τον κώδικα δεοντολογίας, γιατί κάθε υπάλληλος εδώ δεν μπορεί να κάνει τα πάντα όταν έχει εκλογές στις χώρες του και όταν είναι υποψήφοι κοιτάμε πόσο καιρό δουλεύει όντως εδώ ή πόσο καιρό περνάει στην προεκλογική του εκστρατεία. Αντί να είναι εδώ και να δουλεύει για μας. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον εισηγητή, τον κύριο Λιντεράσκη, έτσι αυτό το ξέχασα. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Θέλω λοιπόν να ξέρω, ο κώδικας δεοντολογίας των υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ενημερωμένος και ελέγχουμε ε, την απουσία του υπαλλήλου ο οποίος είναι υποψήφιος για πολιτικά καθήκοντα στη χώρα του. Ε, του, ε, θέλετε να το η κυρία Γκρέσλη, σε αυτό που είπε η κυρία Ματιέ. Κοιτάξτε, ε, θα ήθελα να στηρίξω απόλυτα αυτά που λέει η κυρία Ματιό. Γιατί με τα χρήματα σε μετρητά παραβιάζουμε την κοινοτική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ξέπλυμα ε, βρώμικου χρήματος. Υπάρχει ένα ανώτατο όριο ε, στα μετρητά που μπορούν να διακινούνται. Άρα δηλαδή πρέπει να σταματήσει αυτό. Και θέλω επίσης να επισημάνω ότι υπάρχει και εσωτερικός έλεγχος επ' αυτού. Σε αυτό τον εσωτερικό έλεγχο αναφέρεται ότι οι συνάδελφοι ε, δίνουν στους ε, βοηθούς ε, πολλά μετρητά. Κοιτάξτε, πρέπει να είναι κανείς ανόητος για να βάζει τη ζωή του σε τόσο μεγάλο κίνδυνο. Απλά και μόνο το να προκαλείται αυτή η εντύπωση και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Γι' αυτό λοιπόν, στην κύριε Λιμπεράτσκι, είναι πολύ σημαντικό το Προεδρείο να λάβει απόφαση και να αλλάξει τον κανονισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκάθαρη η τοποθέτηση σας επί του θέματος, λέει ο Πρόεδρος. Ε, επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, έτσι και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαίρετη εκθεσή του. Η έκθεση αυτή, έτσι κι αλλιώς, έχει να κάνει με το παρελθόν. Η εισηγητή γραμματές ε, του επόμενου προπολογισμού του Κοινοβουλίου είναι κάτι που με απασχολεί εμένα πιο πολύ. Νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμο να κοιτάμε μπροστά παρά πίσω. Πιο πολύ πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για τον προπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Αλλά πολλά από αυτά εξαρτώνται και από αυτά που κάνουμε εμείς τώρα. Οι συνάδελφοι ψήφισαν τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προηγισμό στην προηγούμενη Ολομέλεια. Και υπήρχε εκεί μία παράγραφος η οποία λέει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν νέα κτίρια κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής. Συμφωνήσαμε με αυτό. Για το ΚΑΤ, μάλιστα, ζητήσαμε ενημέρωση όσον αφορά το κόστος του κτηρίου αυτού που έχουμε στο Λουξεμβούργο. Όσον αφορά τώρα τον οίκο της ιστορίας, και εδώ θα ήθελα κάποια ενημέρωση. Έχουμε επιμείνει σε μία παράγραφο να ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις και να δούμε την συγχρηματοδότηση, δηλαδή και η Επιτροπή να συνεισφέρει όσον αφορά το κόστος του κτηρίου αλλά και την διαχείριση του οίκου αυτού ιστορίας. Ορισμένοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στα ταξιδιωτικά έξοδα. Στις κατευθυντήριες γραμμές λέμε ότι πρέπει να αναθεωρηθούν τα ταξιδιωτικά έξοδα και ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το κάνει. Περιμένουμε λοιπόν την ενημέρωσή του μέσα σε επόμενες εβδομάδες. Επίσης υπήρχε και μια παράγραφος όσον αφορά για την εξοικονόμηση από αντιπροσωπείες και εκεί θα υπάρξουν εξοικονομήσει. Τώρα για τον επόμενο προπολογισμό ζητήσαμε πάγωμα σε πραγματικού όρου. κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε αλλαγέ όσον αφορά την εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την μετάφραση και τη διερμηνία, για παράδειγμα. Αν θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, οι συνάδελφοι θα πρέπει να δεχτούν να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε σε ορισμένες περιπτώσεις τουλάχιστον. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε εισηγητά μου για όλα τις συγκεκριμένες συστάσεις που κάνατε. Για όλα αυτά που ελέγχθησαν για την πολιτική ακινήτων ε, δημιουργείται μια πολύ περίεργη εικόνα ε, το να δίνει κανείς μετρητά ε, στις ομάδες επισκεπτών. Και θέλω να αναφέρω κάτι το οποίο θεωρώ σημαντικό. Υπάρχουν όρια υπάρχουν όρια ε, στο πόσα χρήματα μπορούμε να εξοικονομήσουμε. Βεβαίως και να εξοικονομούμε χρήματα, αλλά ε, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και διαρθρωτικά προβλήματα. Ε, το Κοινοβούλιο έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που εργάζεται. Ας μην ξεχνάμε αυτό το τσίρκο, το τσίρκο που γίνεται κάθε μήνα, Βρυξέλλες, πήγαινε έλα. Επίσης, οι εβδομάδες ε, των ε, συνεδριάσεων, πόσο συχνά ε, γίνονται οι συνεδριάσεις και πόσες πολλές συνεδριάσεις συμπίπτουν μέσα σε μία εβδομάδα. Υπάρχει ας πούμε κάποιος κανονισμός που να λέει ότι πρέπει το χρόνο να έχουμε μέχρι και 40 συνεδριάσεις. Υπάρχει κάπου αυτό σε γραπτή μορφή. Μήπως λοιπόν η εργασία στο Κοινοβούλιο πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε κάθε μήνα να υπάρχει και μία τυρκουάζ εβδομάδα έτσι ώστε οι ευρωβουλευτές να κάθονται σπίτι τους και να προετοιμάζονται ή αν θέλετε να ε, μας δίνετε έγκαιρα τα έγγραφα για να ξέρουμε γιατί πράγμα ε, θα κουβεντιάσουμε στις συνεδρίες. Αυτό που θέλουμε επίσης είναι να έχουμε περισσότερο χρόνο για τους ε, εκλογείς μας. Μετά, οι τηλεδιασκέψεις για να αποφεύγονται τα πολλά ταξίδια. Μπορούν να γίνονται περισσότερες τηλεδιασκέψεις. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά διαρθρωτικής φύσεως προβλήματα που μπορούμε να συζητήσουμε ε, και ίσως ε, αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε. Ίσως λοιπόν την επόμενη εβδομάδα μπορούμε να έχουμε μια ενδελεχέστερη συζήτηση ε, επ' αυτού του θέματος να δούμε το θέμα ε, κάτω από άλλο πρίσμα διαρθρωτικό. Βεβαίω έχοντα κατά νου την εξοικονόμηση. Δεν μπορούμε βέβαια να καταργήσουμε τη δημοκρατία επειδή θέλουμε να κάνουμε οικονομίε, αλλά και κάθε οργανισμός έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για συνεδριάσει. Υπάρχει μια τάση μέσα σε μια εβδομάδα να ε, διοργανώνται όλο και περισσότερες ε, συνεδριάσεις, να συμπίπτουν αυτές. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι τι ακριβώς επιθυμούμε, ποιες είναι οι προτεραιότητές μας και ποια είναι τα όρια. Αυτή τη συζήτηση τη θεωρώ σημαντική για λόγους πολιτικούς αλλά και οικονομικούς. Και για άλλη μια φορά ευχαριστούμε θερμά τον εισηγητή και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να γίνει κάποια στιγμή αυτή η ουσιαστική συζήτηση. Ευχαριστούμε κύριε Ζίντεκαρτ ε, Πριν από τον εισηγητή θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Ήτελε. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ τον εισηγητή κύριο Λιμπεράσκη πρώτα απ' όλα για την εξαίρετη εκθεσή του. Έχω δουλέψει και εγώ πάνω σε αυτό το θέμα και ξέρω τι σημαίνει. Πολλά θέματα αναφέρονται στην έκθεση αυτή που ίσως οικονομικά να μην είναι τόσο σημαντικά αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την φήμη του Κοινοβουλίου μας. Ιδιαίτερα στους καιρούς του σημερινούς που ζούμε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν έχω πολύ χρόνο, γι' αυτό εγώ θα αναφερθώ μόνο στο θέμα της ασφάλειας. Έχουμε πάρει πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις εδώ και στην Ολομέλεια. Ελπίζω να τηρηθούν οι αποφάσεις αυτές, να τεθούν σε εφαρμογή δηλαδή. Κοιτάξτε, αυτή είναι η τελευταία μου πολιτική ομιλία εδώ στην Επιτροπή αυτή. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους αλλά και την Γραμματεία για την καλή συνεργασία που είχαμε μαζί. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία ε, σήμερα κάθομαι εδώ, αλλά από αύριο θα κάθομαι πίσω-πίσω. Έτσι είναι τα πράγματα, τι να κάνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάντως για την τόσο καλή συνεργασία που είχαμε. Θα ξαναβρεθούμε βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε Ιτελέ. Ε, με την ιδιότητά μου του Προέδρου αυτής της Επιτροπής ε, και εγώ φρέσκος είμαι αλλά φαντάζομαι ότι εξ ονόματος όλων των συναδέλφων ε, μπορώ να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή την αγαστή συνεργασία που είχαμε κατά το παρελθόν. Σας εύχομαι καλή επιτυχία τη νέα σας ιδιότητα και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η πολύ καλή συνεργασία. Ε, καλή τύχη και ευχαριστούμε και πάλι για τη συνεργασία. Υπάρχει τίποτα άλλο. Η κυρία Γκρέσλε. Βεβαίω, ε, εκ μέρου ε, του ΕΛΚ θα ήθελα να ευχηθώ στον κύριο Ήταλα, καλή τύχη. Να μην ξεχάσεις όμως από πού προέρχεσαι και ε, που θα πας τώρα στο ελεγκτικό συνέδριο. Ε, σου εύχομαι καλή τύχη. Ο κύριος Φαζάκας που και αυτός θα πάει στο ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για μας αλλά και για το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, και χαίρομαι Βίλη για την συνεργασία που θα έχουμε, θα έχουμε στο μέλλον. Η κυρία Αιάλα Σέντερς. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να συμφωνήσω με τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες προς τον κύριο Ιταλά. Είναι αλήθεια ότι θα μας λείψει. Είναι ένας ε, συνάδελφος ε, που ξέρει πολύ καλά να δουλεύει, έχει δείξει μεγάλη πίστη στην ε, Επιτροπή αυτή και έχει δουλέψει αμερόληπτα ε, πάνω στις αρχές του. Φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα βρεθεί από την άλλη πλευρά, γιατί το λεκτικό συνέδριο δίχως άλλο αποκτά ένα πολύ σημαντικό μέλο Και έτσι θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Ό,τι καλύτερο λοιπόν σας εύχομαι και ευχαριστώ και εγώ για την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μα. Άλλος κανείς, όχι, για αυτό το θέμα. Και γι' αυτό λοιπόν δίνω το λόγο για να κλείσει το θέμα ο συνάλφος κύριος ε, Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πράγματι θίγησαν πάρα πολλά θέματα. Δεν μπορώ βέβαια να απαντήσω σε όλα. Ας ξεκινήσω με αυτά που είπε ο κύριος Ήταλα. Πρόκειται δηλαδή για το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως αυτό γίνεται αντιληπτό από την κοινή γνώμη. Και χαίρομαι που ετέθη το θέμα αυτό. Η κυρία Γκρέσλε έθιξε πολλά θέματα που είναι σημαντικά. Εγώ συμφωνώ με όλα. Επιτρέψτε μου καταρχήν να κάνω κάποιες γενικής φύσεως παρατηρήσεις. Εμείς χορηγούμε την απαλλαγή για το 2010. Τώρα βρισκόμαστε στο 2012. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να περιοριστούμε στο έτος 2010. Ετέθησαν κάποια σημαντικά θέματα. Ε, Παραδείγματο χάρη ε, η ε, ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και κρατικών προμηθειών. Πράγματι έχουν γίνει ε, κάποια σημαντικά βήματα και στις, ε, στους κανονικούς και στους έκτακτους διαγωνισμούς. Ή αν θέλετε, ε, η, τα ταξίδια, αυτά αναφέρονται στο 37 και το 38. Πολύ συχνά ισχύει το εξής. Η σύνθεση της αντιπροσωπείας ε, ε, γνωστοποιείται λίγες μέρες ε, πριν από το ταξίδι ή κάποιοι βουλευτές αποσύρονται λίγο πριν από το ταξίδι. θα πρέπει ε, να υπάρχει κάποια, να είμαστε προσεκτικοί. Όταν λένε ότι θα πάνε 7 βουλευτέ, να πάνε τελικά 7 και όχι 3. Εμείς οι ίδιοι οφείλουμε να προσέχουμε. Ή οι ομάδε επισκεπτών. Αυτό είναι ένα θέμα, φλέγον θέμα. Το 2009 Είχαμε κάποιες προτάσεις για τις ομάδες επισκεπτών και εισήχθησαν νέοι κανόνες. Ισχύουν λοιπόν τώρα νέοι κανόνες να δούμε πώς θα λειτουργήσουν αυτοί και μετά ε, να τοποθετηθούμε κατόπιν το δημογραφικό στοιχείο ετέθη αυτό ε, και από την κυρία Κρέσλε και από την κυρία Αγιάλα Σέντα. Πράγματι, οι μισθοί ε, στο Κοινοβούλιο και στο, στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν δεν έχουν καμία σχέση με τους μισθούς ε, που καταβάλλονται στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο. Και εγώ ίδιος ε, το διαπίστωσα αυτό μόνος μου έχω κάνει και εγώ μόνος μου την ε, ε, εμπειρία όσον αφορά τους υψηλόβαθμους και τους ε, χαμηλόβαθμους κατόπιν όσον αφορά για την εξοικονόμηση κονδυλίων. Έγινε λόγος για το κύρος μας, για την εικόνα που δίνουμε προς τα έξω. Ε, επίσης αναφέρθηκε ότι ένα μεγάλο τμήμα των δαπανών ε, αυτές υλοποιήθηκαν όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ο εξωτερικός ορκωτός λογιστής διαπίστωσαν ότι ε, δεν υπήρχαν προβλήματα με αυτές τις ε, δαπάνες. Ο κ. Χάρτουγκ αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ε, έθιξε το θέμα της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων. Πάντως για μας, για τις υπηρεσίες διερμηνίας και μετάφρασης, πράγματι εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πολλές φορές το 60% των συνεδριάσεων αναβάλλονται. Εμείς ε, λοιπόν ε, οι βουλευτές ε, είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να ρυθμίζουμε το ρυθμό της εργασίας μας. Ε, θα ήθελα αυτό να ληφθεί υπόψη. Απαντώ τώρα στον ε, συνάδελφο κύριο ε, Γκεμπράντι. Στην παράγραφο 23 αλλά και στην 25 αναφέρονται τα νέα σημεία της έκθεσης και εκεί απαντούμε στις συστάσεις του 2009. Σε πάρα πολλά σημεία της έκθεσης μιλάμε και για τον προϋπολογισμό του 2011. Άρα δηλαδή διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια στον ε, προϋπολογισμό. Ε, σαφώς και μελετάμε και το τι έγινε το 2009 και το ποιες είναι οι προβλέψεις, οι προβλέψεις για το 2011. Είναι σαφές ότι τα γραφεία ενημέρωσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οφείλουμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητά τους. Ο κύριος Μπαλτσίτης μίλησε για ένα σημαντικό θέμα, ε, για τις, ε, τους χώρους εργασίας, Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες, ε, Στρασβούργο. Πολύ συχνά μιλάμε για το κόστος που προκαλεί το Στρασβούργο, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι η νομοθετική βάση και γνωρίζουμε ότι η διοίκηση του Κοινοβουλίου εργάζεται στο Λουξεμβούργο ο δικός μας ο θεσμός, το Κοινοβούλιο, είναι οργανωμένο με αυτόν τον τρόπο. Ε, διαρωτώμεθα κατά πόσον αυτό πρέπει να είναι έτσι, αλλά κοιτάξτε, δεν είναι κατάλληλη στιγμή να γίνει αυτή η συζήτηση στο πλαίσιο μιας απαλλαγής, αλλά σε άλλο επίπεδο. Ο συνάδελφος κύριος ε, Σόνικ έδειξε και αυτός ε, αρκετά θέματα. Μίλησα με το Γενικό Γραμματέα, τον ε, κύριο Βέλε και ε, είπα ότι η κατάσταση δεν με ικανοποιεί όσον αφορά την επιστροφή ε, των ε, δαπανών. Οι ευρωβουλευτές αντιμετωπίζονται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή πρώτα πρέπει να περιμένουμε ουρά ε, έξω από μια πόρτα και μετά πρέπει ε, να ε, περασπιστούμε τον εαυτό μας και να πούμε ότι δεν κλέψαμε τίποτα. Αυτό είναι ένα θέμα που σίγουρα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της απαλλαγής. Η συνάδελφος κυρία Ματιού, μίλησε για τα ταξίδια 5.000 ευρώ επί 40 και ο, ή μάλλον διά του 40, ο καθένας παίρνει κάποια χρήματα που τα έχει στην τσέπη του. Αναφέρομαι στους επισκέπτες που πρέπει να πληρώσουν το ξενοδοχείο, ε, το εστιατόριο. Τέλος πάντων, το Κοινοβούλιο εξετάζει το θέμα και προσπαθεί να βρει ένα αποτελεσματικότερο τρόπο. Όσον αφορά τον κώδικα τοντολογίας, αναφέρομαι ε, στον κύριο Ντί. Αυτό δεν εντάσσεται που είπατε μέσα στην διαδικασία της ε, απαλλαγής. Ο συνάλφος κύριος Βόγκαν μίλησε για την πολιτική ακινήτων, για τα κτίρια μας. Αυτά που είπατε τα άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Ίσως πρέπει να κουβεντιάσουμε για το θέμα αυτό. Ο συνάδελφος ή συνάδελφος Αγιάλα Σέντερ εξεπλάγει, είπε ότι υπάρχει ε, λιγότερη ασφάλεια. Όχι, κοιτάξτε, τα κονδύλια που διατίθενται για την ασφάλεια είναι ακριβώ τα ίδια. Τώρα μπορεί να άλλαξε η ε, φιλοσοφία. Μέχρι τώρα ε, είχαμε ανάθεση σε τρίτους, Υπήρξαν ε, βέβαια κλοπές, ε, η Γενική Διεύθυνση έχει αλλάξει λιγάκι τη φιλοσοφία της ε, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν στο Κοινοβούλιο όλοι αυτοί που φορούν τις στολές, αλλά πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη για να περιοριστεί ε, και περιοριστεί η ανάθεση έργων σε τρίτους. Κατόπιν, υπάρχουν ε, διαμαρτυρίες, ε, γνωρίζουμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ε, ασφάλεια μέσα στο κτιριό μας. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν και θα σας δοθεί ευκαιρία να καταθέσετε τροπολογίες μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές ε, προτιθέμεθα να ολοκληρώσουμε τις ε, εργασίες μας ε, και κατά τα άλλα βεβαίως και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λιμπεράτσκι. Η προθεσμία, η διορία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 5η Μαρτίου, 12 η ώρα και μετά η απόφαση θα ληφθεί στις 26-27 Μαρτίου του 2012. Μήπως ε, μπορείτε την ε, διορία να την μεταθέσετε σε 6 ώρα το απόγευμα, γιατί 12 η ώρα ε, το πρωί της Δευτέρας δεν σημαίνει τίποτα. Είτε Παρασκευή είτε Πέμπτη αν θέλετε. Θα δούμε, θα προσπαθήσουμε, θα το δει η Γραμματεία για να δούμε κατά πόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό και θα σας ενημερώσουμε. Ε, γιατί αλλιώς ε, θα είμαστε υπό τεράστια πίεση αν δεν αλλάξετε τη διορία. Ε, πρόεδρος, πράγματι θα το προσπαθήσουμε για αυτή την έκθεση γιατί είναι πολύ σημαντική να μεταθέσουμε τη διορία κατάθεση τροπολογιών στις 6 ώρα το απόγευμα. Κατόπιν τούτου κλείνει η συζήτηση για αυτό το θέμα της σημερινής διάταξης και πάμε στο επόμενο που αφορά στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Και εδώ πρόκειται για τους κανόνες. Ε, ο κύριος Γόβεν από το ε, ε, ελεγκτικό συνέδριο είναι ο εισηγητής μας. Η κύριο Φαζάκας, τους καλωσορίζω, τους κυρίους Φαζάκας και Μισελ Κρετίν. Και θα ήθελα να πω ότι ξεκινώντας θα ακούσουμε την τοποθέτηση του ελεγκτικού συνεδρίου. Μετά θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή μας. Σε ποιον θα δώσω παρακαλώ το λόγο από το ελεγκτικό συνέδριο. Παρακαλώ κύριε Φαζάκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω με την ε, έκθεση, επιτρέψτε μου να σας ε, συγχαρώ ε, για την την εκλεγή σας, τον διορισμό σας σε αυτή τη θέση. Εγώ ε, υπήρξα στη θέση αυτή, ε, γνωρίζω πόσο σημαντική είναι, σας εύχομαι <clears throat> καλή τύχη, υπομονή και καλή επιτυχία. Και εφόσον ε, είμαι στα συγχαρητήρια, συγχαίρω και τον κύριο Ιτάλα ο οποίος είναι το νέο μέλος ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Χαιρόμαστε ε, για την εκλογή του ε, και πρέπει, θέλω να αποσχεθώ στην κυρία Γκρέσλα ότι όχι μόνο θα του φερθούμε φιλικά αλλά και θα προσπαθήσουμε να ε, ικανοποιήσουμε όλες τις αιτιολογημένες επιθυμίες της όσον αφορά στο ελεκτικό συνέδριο. Τώρα θα στραφώ προς τα αγγλικά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, καταρχάς σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου για τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Ταμείων για την περίοδο 14 με 20. Πριν επισέλθω στις λεπτομέρειες θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή σας κύριο Ντέρεκ Βόγκαν για την εξαιρετική ποιότητα της δουλειάς του. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για το πνεύμα συνεργασίας του γιατί οι επαφές που είχαμε ήταν πολύ χρήσιμες και για τις δύο πλευρές. Οι συζητήσεις μας έδειξαν ότι η γνωμοδότηση του συνεδρίου συμφωνεί με την προσέγγιση και τη δική σας. Και η συμφωνία αυτή ενδυναμώθηκε και από την θέληση του κυρίου Βόγκαν να συμπεριλάβει ορισμένες από τις συστάσεις μας. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να υπενθυμίσω ότι το σχέδιο κανονισμού προβλέπει, ε, θέτει ορισμένα πολιτικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν από παλιτικούς, δηλαδή τον δημοκρατικά, τα δημοκρατικά εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό στη γνωμοδότησή του το ελεκτικό συνέδριο δεν θέλησε ούτε να υποστηρίξει ούτε να καταδικάσει καμία πρόταση του σχεδίου κανονισμού διότι εσείς οι νομοθέτες πρέπει να αποφασίσετε αν γίνονται αποδεκτές οι προτάσεις ή όχι. Το συνέδριο θεωρεί ότι έχει συμβουλευτικό ρόλο ως προς τις επιπτώσεις και τα υπέρ και τα κατά των προτάσεων με τα συμπεράσματά του και τις συστάσεις του. Άρα είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σας με αυτήν την ε, συμφωνία μας δείχνει ποια ακριβώς είναι τα τεχνικά προβλήματα που ακόμη εκκρεμούν. Παρουσιάζοντας τη γνωμοδότησή μας θα ήθελα να πάω παράγραφο με την παράγραφο και να σας συζητήσω σημείο προς σημείο τα συμπεράσματα. Ξέρω όμως ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο και γι' αυτό δεν θα το πράξω. Δεν θα το πράξω. Θα ήθελα λοιπόν να περιοριστώ σε τέσσερα μόνο βασικά θέματα και σε τρία συγκεκριμένα σημεία για τη διαχείριση. Πρώτον, το θέμα των δαπανών που θα ήταν μια ευκαιρία της προστιθέμενης αξίας των μέτρων της Ένωσης. Έχουμε προτείνει να αλλάξουν οι δαπάνες για να είναι πιο αποδεκτές με βάση συγκεκριμένα σχέδια και αποζημιώσεις που να βασίζονται σε αποτελέσματα. Παρά όμως αυτή την έμφαση στα αποτελέσματα το προτινόμενο πλαίσιο για την περίοδο 14-20 παραμένει βασιζόμενο στο input και στη διαχείριση μάλλον παρά στα αποτελέσματα. Εκτός αυτού, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο μπορεί να δαπανηθεί σε υπερβολικά πολλές δραστηριότητες και γι' αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να καθοριστεί μια κρίσιμη μάζα που να επιτρέπει παρεμβάσεις της Ένωσης με απτά αποτελέσματα. Οι όροι που τίθενται εξάντε είναι ένα βασικό στοιχείο που θα μπορούσε να ενδυναμώσει την λογική της παρέμβασης των ε, αντιδράσεων της Ένωσης διευκολύνοντας τα πράγματα και γι' αυτό νομίζουμε ότι τα κονδύλια που προτείνονται για την έρευνα και την καινοτομία είναι κάτι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Πολλές πτυχές των ε, διακανονισμών που προτείνει η Κομισιόν προβλέπονται για δεύτερη φάση. Ιδιαίτερα το, τα όσα προτείνονται για τη συνοχή. Μπορεί όλα αυτά να ξεπερνούν τα συγκεκριμένα θέματα που έχουν προβλεφθεί και να έχουν επιπτώσεις και για άλλα τους τομείς της νομοθεσίας. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να διασφαλιστεί η συνοχή και συνέπεια μεταξύ των διαφόρων λεπτομεριών και στο σύνολο των κοινών κανόνων. Άρα είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε την αναγκαιότητα που υπάρχει να διασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ του Common Provisions Regulation και του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Αλλά εσείς θα κρίνετε βέβαια, γιατί είστε πιο αρμόδιοι από μένα. Η προτινόμενη μείωση των εθνικών πληρωμών καθώς και η εφαρμογή των όρων που προτείνονται για τα μακροοικονομικά πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά για να μην υπάρξουν αντιπαραγωγικά αποτελέσματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πληροφορήσω ότι τη Δευτέρα στην Επιτροπή Περιφερειών είχαμε συζητήσει την κατάσταση λεπτομεριακώς και χάρηκα ιδιαίτερα γιατί είδα ότι η γραμμή των εισηγητών σας συμφωνούν απόλυτα με, με τα αποτελέσματά μας. Ελπίζω λοιπόν ότι μετά από τις συζητήσεις αυτές μπορεί να δεχτείτε τις συστάσεις μας και στην έκθεσή σας. Έρχομαι τώρα στο θέμα της διαχείρισης. Θα ήθελα να τονίσω τα εξής τρία θέματα. Οι διακανονισμοί για τη δαπάνηση των κονδυλίων συνοχής παραμένουν πολύπλοκοι και πρέπει να μειωθεί το διοικητικό άχθος που αντιμετωπίζουν όσοι ωφελούνται από αυτά τα κονδύλια. Το έγγραφο εργασίας σας λέει σωστά ότι η απλοποίηση πρέπει να γίνει τεχνιέντος, δηλαδή να αποφευχθεί το άχρηστο διοικητικό άχθος, ενώ θα υπάρχει εγγύηση του ελέγχου χωρίς όμως μεγάλη πολυπλοκότητα των κανόνων. Επίσης πρέπει να υποθεί ρητά ότι οι προτινόμενες αλλαγές στοχεύουν στην επίτευξη των απλοποιήσεων υπέρ όσων ωφελούνται από τα ταμεία. Γιατί πολλές φορές δημιουργείται άχρηστος φόρτος εργασίας για την Ένωση και τις εθνικές διοικήσεις. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να προετοιμαστούν καταλήλως και με τους κατάλληλους πόρους. Ο προτινόμενος κανονισμός προ, ε, στοχεύει στο συντονισμό της εφαρμογής και της δαπάνησης μεγάλου αριθμού ταμείων. Πρέπει βέβαια τα ταμεία αυτά να δαπανηθούν όπως πρέπει ώστε να στηρίζουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Και για να επιτευχθούν αυτοί οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, τα συστήματα εφαρμογής και ελέγχου πρέπει να είναι αποτελεσματικά από την αρχή. Αποτελεσματική εποπτεία δηλαδή και λογοδοσία από την Επιτροπή για τη χρήση των κονδυλίων θα ήταν κάτι το βασικό. Επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο της ε, ανεπαρκούς εποπτείας που μπορεί να οδηγήσει τελικά στον πολλαπλασιασμό των ελέγχων. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι δημοσιονομικοί διορθωτικοί μηχανισμοί θα αντισταθμίσουν επαρκώς τα πιθανά λάθη και ότι όλα τα υλικά προβλήματα θα λυθούν από την αρχή. Αυτό σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα της εθνικής διαχείρισης πρέπει να διασφαλίζεται από την αρχή. Όπως σωστά λέει και το έγγραφο εργασίας σας, ένα σωστός έλεγχος ιδιαίτερα μέσω του ελέγχου διαπιστευτηρίων που θα κάνει η Κομισιόν θα διευκολύνει την λύση των προβλημάτων για την αποφυγή άχρηστων δημοσιονομικών διορθώσεων. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι οι διαπιστώσεις του εξαιρετικού εγγράφου εργασίας σας και της γνωμοδότησης του ελεγκτικού συνεδρίου συμφωνούν μεταξύ τους. Ελπίζω στο έγγραφο εργασίας σας να λάβετε υπόψη σας και τις προτάσεις μας και επομένως τελικά στον τελικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, θα ήθελα να ζητήσω από τον συνάδελφό μου και συνεισηγητή της γνωμοδότης, τον κύριο Μιχαήλ Κρετέν, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φαζάκα, για τόσα μας είπατε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μισελ Κρετά, τον συναδελφό σας. Παρακαλώ. Δεν εδώ. Α, όχι τώρα. Δεν θα πάρει το λόγο τώρα. Καλώς. Α, όχι. Θα μιλήσει παρόλα αυτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να προσθέσω δύο παρατηρήσεις μόνο στο όσα είπε ο συνάδελφός μου, ο κύριος Φαζάκας. Η πρώτη μου παρατήρηση έχει να κάνει με το εξή. Όπως γνωρίζετε, ε, το Ταμείο για την ε, ε, Ανάπτυξη της Υπέθρου και εκείνο για την Αλία συμπεριλαμβάνονται στις κοινέ διατάξεις του σχεδίου κανονισμού που εξετάζεται σήμερα. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι η συμπερίληψη αυτών των δύο ταμείων έχει ως στόχο να καθαρίσει μια κοινή στάση για τα πέντε ταμεία τα οποία καλύπτονται από το σχέδιο κανονισμού, δηλαδή τα τρία διαφορετικά ταμεία και τα δύο ταμεία που έχουν να κάνουν με τους φυσικούς σπόρους. Όμως, το ελεγκτικό συνέδριο σκέφτηκε ότι παρόλα αυτά υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την αρχή διαχείρισης των κονδυλίων αυτών, χωρίς να αιτιολογούνται αυτές όμως οι διαφορές. Και θα σας δώσω κάποια παραδείγματα όσον αφορά τους κανόνες διαχείρισης των ταμείων. Πρώτο λοιπόν παράδειγμα έχει να κάνει με την εκαθάριση των λογαριασμών. Αυτό εξάλλου είναι ένα θέμα το οποίο ο εισηγητής σας το σημειώνει πάρα πολύ καλά. Το σύστημα λοιπόν αυτό το οποίο προβλέπεται για το Κοινωνικό Ταμείο, για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για το Ταμείο Συνοχής είναι διαφορετικό από το σύστημα καθάρισης λογαριασμών το οποίο ισχύει για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Για την ανάπτυξη της υπαίθρου το σύστημα καθάρισης λογαριασμών καλύπτει και την αξιοπιστία των λογαριασμών όπως υποβάλλουν οι διάφορες, διάφοροι οργανισμοί και την νομιμότητα και κανονικότητα των ε, δράσεων έτσι όπως αναφέρονται στους λογαριασμούς. Ενώ αντίθετα για τα διαρθρωτικά ταμεία η εκαθάριση λογαριασμών δεν καλύπτει παρά μόνο τη δημοσιονομική ετήσια εκαθάριση, την αξιοπιστία δηλαδή των λογαριασμών και δεν καλύπτει την νομιμότητα και κανονικότητα των ε, δράσεων. Δεν έχουμε καταλάβει γιατί υπάρχει η διαφορά αυτή. Μάλιστα, δεδομένου ότι το θέμα της κανονικότητας και νομιμότητας όσον αφορά τα διευθυντικά ταμεία εξετάζονται σε διαφορετικό κεφάλαιο του σχεδίου κανονισμού. Ένα δεύτερο παράδειγμα διαφοράς μεταχείρισης που είναι αδικαιολόγητη κατά τη γνώμη μας είναι το εξή. Στην περίπτωση των διαρθρωτικών ταμείων, όταν η Κομισιόν επιβάλλει μία ε, δημοσιονομική διόρθωση για να επιβάλλει κυρώσεις την μη κανονική, μη νόμιμη διαχείριση των κονδυλίων, τότε η διάταξη, μάλλον ε, αυτό στον οποίο εφαρμόζεται αυτό, μπορεί, έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι πρόκειται για ένα ποσό χαμηλότερο από την εκτίμηση στην οποία κατέληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε η διόρθωση αυτή η πιο χαμηλή τελικά ισχύει. Όμως αυτή η δυνατότητα ένστασης όσον αφορά τα ποσά ε, ανάκτησης μετά από τις δημοσιονομικές διορθώσεις δεν ισχύει στην περίπτωση της γεωργίας και των φυσικών πόρων. Και εδώ λοιπόν η απορία μας είναι γιατί να υπάρχει αυτή η διαφορετική μεταχείριση. Έρχομαι τώρα στη δεύτερη παρατήρησή μου. Αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι το σχέδιο κανονισμού όσον αφορά τα διευθυντικά ταμεία εισάγει ένα σύστημα το οποίο ήδη ισχύει για τα γεωργικά ταμεία. Το σύστημα αυτό συνίσταται στο να υπάρχει διαπίστευση από τα κράτη-μέλη σε εθνικούς οργανισμούς οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών δαπανών. Το Ελεκτικό συνέδριο λοιπόν πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι και ο τελικός υπεύθυνος για την εκτέλεση του προπολογισμού το συνέδριο λοιπόν πιστεύει ότι η Κομισιόν πρέπει να επιβεβαιώνει στην αρχή κάθε δημοσιονομικής περίοδου ότι οι εθνικοί οργανισμοί ελέγχου ε, που έχει διαπιστεύσει το κάθε κράτος μέλος πράγματι είναι σε θέση να φέρουν σε πέρα στα καθήκοντά τους. Ε, δεν προβλέπεται όμως μια τέτοια επιβεβαίωση στο σχέδιο κανονισμού προς το παρόν. Αν όμως εισαχθεί, τότε η Κομισιόν θα είναι πολύ περισσότερο σε θέση να βασιστεί στις εργασίες αυτών των οργανισμών διαχείρισης και ελέγχου, κάτι το οποίο επί του παρόντος δεν ισχύει. Το τελευταίο που έχω να πω όσον αφορά τη διαχείριση των διορθωτικών ταμείων είναι το εξή. Το σχέδιο κανονισμού δεν προβλέπει την διαπίστευση εθνικών οργάνων ε, λογιστικού ελέγχου το σχέδιο κανονισμού περιορίζεται στην εξή πρόβλεψη. Λέει ότι το κράτος μέλος ορίζει ποια θα είναι η αρχή ελέγχου, χωρίς όμως σύστημα διαπίστευσης. Και εδώ λοιπόν, δεδομένου ότι η Κομισιόν είναι ο κύριος χρήστης των ε, εργασιών αυτών των εθνικών οργάνων ελέγχου, λογιστικού ελέγχου, το συνέδριο πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιβεβαιώνει την ποιότητα των συστημάτων και την αξιοπιστία των εθνικών αυτών αρχών λογιστικού ελέγχου. Εξάλλου, έχω διαπιστώσει ότι ο συγητή σα και αυτός προτείνει το ίδιο πράγμα όπως και το λεκτικό συνέδριο. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου λοιπόν κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας τις παρουσιάσω. Merci, Monsieur Chrétien. Vielen Ευχαριστούμε πολύ. Ε, νομίζω ότι ε, τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο πρώτος έχει το λόγο συγητής, ο κύριος Βον. Ευχαριστώ και τον κύριο Καζάκας και τον κύριο Κρετέν για τη συμβολή τους και για την ε, γνωμοδότηση που παρουσίασαν. Νομίζω ότι τα δύο μας έγγραφα συμφωνούν εν Στο έγγραφο εργασίας βλέπετε ότι αρχίζουμε μιλώντας με το ρυθμό λάθους. Είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και κάθε χρόνο το τονίζουμε. Είναι κατανοητό αυτό γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα ενωσιακά χρήματα δαπανούνται σωστά. Το λάθος βέβαια δεν είναι και απάτη αναγκαστικά, όταν μιλάμε για αριθμό λάθους δεν ανταποκρίνεται αυτό στο κατά πόσον αποτελεσματικά εκτελούνται τα προγράμματα. Όλοι όμως θα συμφωνούσαν ότι πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την πρόληψη των λαθών και των απατών. Ένα παράδειγμα είναι η ιδέα των διαπιστευτηρίων, δηλαδή να εκαθαρίζονται τα κράτη-μέλη εξάντε από την Κομισιόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο δημοσιονομικός έλεγχος είναι διαφορετικό πράγμα. Αυτά τα διαπιστευτήρια είναι καλή ιδέα και την υποστηρίζουμε, αλλά πρέπει επίσης τελικά η ευθύνη να παραμείνει στην Κομισιόν. Αυτό να τονιστεί ιδιαίτερα. Κάτι άλλο που λέμε κάθε χρόνο στην Επιτροπή μας ως προς την πολιτική συνοχή και τα διαρθρωτικά και άλλα ταμεία είναι η ανάγκη για απλοποίηση. Πάντοτε λέμε ότι μια από τις λύσεις για να μειωθεί ο ρυθμός των λαθών είναι η απλοποίηση των κανόνων. Το λέμε κάθε χρόνο, τώρα πια είναι καιρός να εφαρμοστεί ένας μηχανισμός διαδικασίες που να επιτρέψουν τέτοια απλοποίηση. Μάλιστα η Κομισιόν κάνει μερικές σχετικές συστάσεις και κοινούς κανόνες. Επίσης εκφράζει την ιδέα των flat rate payments ή των καταποκοπήν ποσών. Πρέπει να γνωρίζουμε βέβαια αν θέλουμε να απλοποιηθούν οι κανόνες για όλους τους ωφελούμενους, για τα κράτη-μέλη ή μόνο για τα ενωσιακά όργανα. Αν θέλουμε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και για τους ωφελούμενους, τότε ίσως πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό και τα κράτη-μέλη, και αυτό το λέει η εκθέση του ελεκτικού συνεδρίου. Κάτι άλλο ιδιαίτερα σημαντικό για μας ως προς την επιτοχή συνοχής είναι το θέμα των παγωμάτων και των διακοπών. Αυτές οι διακοπές των πληρωμών έχουμε συζητήσει πολλές φορές αν πρέπει να είναι συστηματικές ή όχι. Εγώ είμαι υπέρ των συστηματικών, αν και μπορεί μερικοί να διαφορούν. Άλλη πρόταση της Κομισιόν είναι να αλλάξουν τα χρονικά περιθώρια από τους έξι μήνες στους εννέα Και με αυτό συμφωνώ. Ο τομέας για τον οποίο χαίρομαι ιδιαίτερα στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ότι καταδικάζει αυτή την ιδέα των όρων, μακροοικονομικών όρων για το μέλλον στην πολιτική συνοχή. Πράγματι πρόκειται για τεράστιο λάθος. Δεν ξέρω αν κανείς μπορεί να μιλήσει υπέρ. Μου φαίνεται ότι είναι λάθος να τιμωρούνται οι περιφέρειες για λάθη κεντρικών κυβερνήσεων. Αν ένα κράτος δημοσιονομικά και οικονομικά έχει πρόβληματα, δεν θα έπρεπε να του αφαιρούμε και τα διαρθρωτικά και περιφερειακά κονδύλια του. Πρέπει η Κομισιόν αυτό να το ξαναδεί. Και χαίρομαι γιατί το νοικτικό Συνέδριο το αναγνωρίζει αυτό. Στο έγγραφο εργασίας τίθενται και άλλα προβλήματα. Ένα είναι οι δηλώσεις διαχείρισης. Πολλές φορές το έχουμε πει και αυτό. και το θέμα μιας ενιαίας εκαθάρισης αντί στο τέλος του κάθε προγράμματος ή περίοδου. Επίσης στο έγγραφο εργασίας μιλάω για το θέμα των δημοσιονομικών διορθώσεων και αυτό είναι θέμα που έχει συζητηθεί πολλές φορές στην Επιτροπή μας. Και η πρόταση της Επιτροπής είναι κάτι που το δέχομαι, δηλαδή η καθαρή μείωση για τα κράτη-μέλη. Είναι κάτι που θα μπορούσε να λύσει τα προβλήματα και να μην πληρώνει δύο φορές ο φορολογούμενος και οι φορολογούμενοι. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία του εγγράφου εργασίας και θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά το ελεγκτικό συνέδριο για τη βοήθειά του. Είναι βέβαια απλώς ένα έγγραφο εργασίας και με χαρά θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους τους επόμενους μήνες, επόμενες εβδομάδες και μήνες Προβλέπεται και στις 23 Απριλίου μια άλλη ανταλλαγή απόψεων και τελική έγκριση στις 30 Απριλίου. Έχουμε λοιπόν λίγο χρόνο. Εν τω μεταξύ θα ήθελα να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνεργασία με τον κύριο Βόν είναι πάρα πολύ καλή. Η συζήτηση γίνεται την κατάλληλη χρονική στιγμή. Ε, για μένα τουλάχιστον αυτό μου φρεσκάρει την όλη προβληματική γιατί αύριο ε, είναι και η τελευταία φάση ε, συζήτησης με το Συμβούλιο για την επιμερισμένη διαχείριση. Και ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Γκάιερ γιατί είναι πάντα παρόν και αυτό το βρίσκω ιδιαίτερα επικοδομητικό. Αυτά τα οποία διαπιστώνει το ελεγκτικό Συνέδριο και γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικά. Και επιτρέψτε μου τώρα να σας πω σύντομα ποιες είναι οι μέχρι τώρα δυσκολίες ε, στις διαπραγματεύσεις σε αυτά που το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί σημαντικά. Πιστοποίηση των εθνικών αρχών ελέγχου στα κράτη-μέλη. Αυτός είναι ένας πραγματικός αγώνας με το Συμβούλιο. Ε, μέχρι τώρα για κανένα άλλο θέμα δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε συμφωνία. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις του Συμβουλίου και ελπίζω αύριο να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα της πιστοποίησης ποια θα είναι η και αυτή είναι η διαμάχη με την Κομισιόν. Ποιο θα είναι ο ρόλο τη Κομισιόν σε όλο αυτό. Ευχαριστώ πολύ το ελεγκτικό συνέδριο που λέει ότι είναι σημαντικό ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εμεί θεωρούμε ότι πρέπει να ορίσουμε αυτό το ρόλο. Γιατί? Διότι δεν επιθυμούμε μετά από δύο-τρία χρόνια να εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το πρόβλημα των διορθώσεων, διότι το σύστημα στήθηκε λάθος από την αρχή. Υπάρχουν λοιπόν τροπολογίες, ε, αυτό το βρίσκω πολύ έξυπνο, λέμε ότι η Κομισιόν ε, θα πρέπει να προχωρήσει με βάση τη δική της την αξιολόγηση κινδύνου ή μετά από αίτημα των κρατών μελών. Και το ότι το απορρίπτει αυτό η Κομισιόν το βρίσκω ιδιαίτερα λυπηρό, γιατί δεν είναι δυνατόν η Κομισιόν να κάθεται ε, άνετα και μετά να λέει ε, θα σας αξιολογήσουμε τώρα, θα σας δώσουμε βαθμούς α, β, θα παίζουμε δηλαδή το ρόλο του διαιτητή. Μα δεν είναι αυτός ο ρόλος της Κομισιόν, ούτε έχει οριστεί με αυτόν τον τρόπο ε, στις συνθήκες. Το Συμβούλιο για πολύ καιρό ε, ήταν απρόσιτο για μεγάλο χρονικό διάστημα το Συμβούλιο δεν επεξεργάστηκε το άρθρο αυτό, διότι είχαν στο εσωτερικό τους πολλές συζητήσεις. Και τέλος, αυτό το οποίο υπέβαλε το Συμβούλιο αφήνει όλα ανοιχτά όλο το οικοδόμημα. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και εμείς αυτό δεν το δεχόμαστε γιατί αυτό σημαίνει ότι απλά συνεχίζονται τα υπάρχοντα προβλήματα. Τώρα, οι προτάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου εν μέρη τις λάβαμε υπόψη μας. Σήμερα τη νύχτα, το βράδυ θα τα δω αυτά έτσι ώστε αύριο το πρωί να είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Το έγγραφο εργασία του συναδέλφου κ. Βον το βρίσκω ιδιαίτερα επικοδομητικό και θα συμμετάσχω με χαρά ε, στις συζητήσεις. Η θέση της Επιτροπής Ελέγχου Προεπολιμών πρέπει πράγματι να οριστεί έγκαιρα. Συμφωνώ ε, με αυτά που είπε ο ε, ορκωτός λογιστής κύριος Κρετέν Δηλαδή η πρόθεση είναι να πλησιάσουν λίγο οι κανονισμοί και αυτό δεν το κατάφερε η Κομισιόν γιατί το κάθε ταμείο επιμένει στα δικά του. Λυπάμαι πάρα πολύ που η προστιθέμενη αξία από την απλούστευση της διοίκησης δεν προκύπτει. Και λυπάμαι πολύ που είμαι αναγκασμένη να πω ότι ως Κοινοβούλιο δεν είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε ένα σύστημα με τροπολογίες, διότι δεν μας δίνει τη δυνατότητα κομισιών. Απλά δεν μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Ε, λυπάμαι λοιπόν πραγματικά πολύ για το ότι δεν προσπαθήσαμε να επιτύχουμε καλύτερη διοίκηση από το πλησίασμα των ταμείων. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση και ίσως μετά το 2020 ε, να επιτύχουμε περισσότερα με άλλους συγητές. Αλλά ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη πολύ σωστά ε, παραπονιούνται για τη γραφειοκρατία. Αυτό που μετράει τώρα είναι το συντομότερο δυνατό να προχωρήσουμε με ικανοποιητικά αποτελέσματα. αποτελέσματα. Συνάλφε κύριε Βόν, ίσως αύριο το βράδυ ε, μπορούμε να σας ε, ανακοινώσουμε τη θέση μας ε, για το άρθρο 56 για την επιμερισμένη διαχείριση. για να ξέρετε περίπου ποια είναι η γνώμη μας για τα συστήματα ελέγχου. Ελπίζω να το κάνουμε αυτό αύριο το βράδυ. Και αν είναι κάποιος εδώ στην αίθουσα από το Συμβούλιο, κάνω έκκληση και αυτοί αύριο το βράδυ να δώσουν τη τους. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, γιατί αλλιώς ε, δεν θα μπορέσουμε πάλι να ενοποιήσουμε τους κανόνες και αυτό θα ήταν μοιραίο για όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γκρέσλε, ε, πολύ μεγάλο ε, πλεονέκτημα το ότι στην Επιτροπή μας έχουμε και την εισηγήτρια της Επιτροπής Προϋπολογισμών για το θέμα αυτό. Άρα δηλαδή, καλό διότι τα θέματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Έχω τώρα ε, το συνάδελφο Οντί που ζήτησε το λόγο, ε, δεν βλέπω να το ζήτησε άλλος, ο κύριος Οντί παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Αναρωτιέμαι, η περίοδος αλλαγής των ε, δημοσιονομικών προοπτικών μέχρι το 2013 και επόμενο πάει μέχρι το 2020, μήπως θα έπρεπε να αξιολογήσουμε γενικότερα την δημοσιονομική μας ε, οργάνωση και να δούμε πόσο κοστίζει. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια δίκη, είτε πρόκειται για τη συλλογή, είτε για την κατανομή πόρων, κοστίζει. Και ο έλεγχος βέβαια. Και όταν μάλιστα βλέπουμε πόσο περίπλοκο είναι το σύστημα αυτό της επιμερισμένης διαχείρισης μέσα στο οποίο βρίσκουμε και τα περισσότερα σφάλματα, ακόμα και αν η κατάσταση βελτιώνεται, αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να αξιολογήσουμε το σύστημα. Το κάνουμε με τις απαλλαγές, με την έκθεση αυτή που είναι καλής ποιότητας θα μπορούσαμε. Οπότε ρωτάω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή να φτιάξει τη δικιά της δημοσιονομική ε, λειτουργία. Τα κράτη-μέλη δεν θέλουν, θέλουν την επιμερισμένη διαχείριση βέβαια. Είναι η λογική του θέλω τα λεφτά μου πίσω, I want my money back. Όμως, όσο περνάει ο καιρός και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά μεγαλύτερη οικονομική, δημοσιονομική και στρατηγική σημασίας ε, ε, διάσταση, δεν θα έπρεπε να έχει τη δικιά της δημοσιονομική λειτουργία. Όπως έχουμε το 20% για την έρευνα κτλ. Πάει καλά και εκεί είναι που έχουμε και χαμηλότερα ποσοστά ασφάλματος. Δεν ξέρω τεχνικά πώς μπορεί να λυθεί το θέμα. Πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, το 2019 δηλαδή, για να το θέσουμε. Εγώ νομίζω όμως μία αξιολόγηση χρειάζεται. Κυρίως θέλω να ξέρω πόσο κοστίζει όλη αυτή η οργάνωση, όλα αυτά τα συστήματα διαχείρισης και λογιστικού ελέγχου στα διάφορα κράτη-μέλη δεν κοστίζουν πάρα πολλά. Eh, eh, Ευχαριστώ. Εγώ αναλαμβάνω τώρα ως πρόεδρος, μια που είχε άλλες ανελημμένες υποχρέωσεις ο πρόεδρος. Οπότε, τώρα θα ακούσουμε κάποια αντίδραση ενδεχομένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ή κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπω θέλει το λόγο εδώ. Εσείς, ναι. Παρακαλώ, πείτε μα και ποιο είσαστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νίκολας Μάρτιν ονομάζομαι και είμαι αναπληρωτή Γενικός Διευθυντή για την Περιφερειακή Πολιτική. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω στην Επιτροπή σας σήμερα και να συμμετάσχω στη συζήτηση αυτή που έχει να κάνει με την γνωμοδότηση του Λεκτικού Συνεδρίου σχετικά με την πρόταση τη Επιτροπής για πέντε τα μία όσον αφορά την νέα δημοσιονομική περίοδο. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι εκτιμούμε όλους ιδιαίτερως ε, την εργασία που επιτελείται στο λεκτικό συνέδριο, όπως επίσης και το έργο του δικού σας εισηγητή. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσε συστάσεις και στη γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου και στο έγγραφο εργασίας, το οποίο ελπίζουμε ε, θα προχωρήσει μετά τις διαπραγματεύσει. Πρώτα απ' όλα θα αναφερθώ στη γνωμοδότηση του Λεκτικού Συνεδρίου. Εκεί υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία στηρίζουν και την πρόταση της Κομισιόν. Βλέπουμε ότι στηρίζεται το θέμα του συντονισμού, ε, το θέμα της αιρεσιμότητας εξάντε, η προσέγγιση επίσης για το ετήσιο κλείσιμο, ε, για το συνδυασμό επίσης διαφόρων στοιχείων αλλά θα έρθω στα ιδιαίτερα θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Φαζάκας, πρώτα απ' όλο. Για το θέμα της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε προχωρήσει σε μια μεγάλη αλλαγή. Ε, τα ταμεία αντί να βασίζονται στο input, πιο πολύ μας ενδιαφέρει να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα. Δηλαδή, έχουμε πολύ περισσότερους δείκτες, ε, τους εντοπίζουμε τους δείκτες αυτούς και έχουμε και μηχανισμούς ε, για να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες εφόσον ε, δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους δείκτες. Υπάρχει ένα σύστημα δηλαδή το οποίο θα αλλάξει πιστεύουμε κατά πολύ τη λογική των παρεμβάσεων που γίνονται από την πολιτική συνοχής προκειμένου να επικεντρωθούμε περισσότερο στα αποτελέσματα για το θέμα ε, των ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων. Εδώ φυσικά και υπάρχουν πολλές που προτείνονται και θα υπάρξουν και περισσότερες λεπτομέρειες. Γίνονται αυτά. Συμφωνούμε ότι όντως πρέπει να υπάρχει πλήρης ε, συμφωνία με τους κανόνες. Γι' αυτό και συζητούμε τα κύρια στοιχεία με τις νομοθετικές αρχές στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων. Επίσης πρέπει να συνάδουμε και με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Το λέμε αυτό στην πρότασή μας. Αλλά και γι' αυτό συνεργαζόμαστε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται βάσει του άρθρου 56 του δημοσιονομικού κανονισμού. Για το θέμα της μακροοικονομικής ερεσιμότητας. Αυτά έχουν να κάνουν με την πρόταση της Επιτροπής για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε με μια ισορροπημένη δημοσιονομική πρόταση. Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις για το κάπινγκ, για τις μειώσεις, εξαρτώνται από τις δυνατότητες των κρατών μελών και πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε ότι υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Πάντως για το θέμα της αρεσιμότητας είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη λογική πίσω από αυτό και μένουμε σε αυτό. Δεν είναι ένα σύστημα που τιμωρεί κανένα. Είναι ένα σύστημα το οποίο ξεκινάει εφόσον συστηματικά κάποιο κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις που κάνει το Συμβούλιο στα πλαίσια των διαδικασιών ε, υπερβολικών ε, ελλημάτων ε, κλπ. Οι επιπτώσεις δεν είναι άμεσες, αλλά υπάρχει κάποια άρση η οποία με τη σειρά της σταματά εφόσον τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν σωστές δράσεις. Τώρα, για το θέμα του ελέγχου της διαχείρισης, πράγμα στο οποίο αναφέρθηκαν και ο κύριος Φαζάκας και ο κύριος Κρετάν και ο κύριος Βον. Η διαπίστευση ήταν ε, ένα βασικό θέμα. Για την ε, πολιτική συνοχής έχει έναν ρόλο η Κομισιόν, προσέγγιση κινδύνου δηλαδή. Και πιστεύουμε ότι έτσι διασφαλίζεται ότι τα συστήματα είναι αποτελεσματικά από την αρχή. Έχει να κάνει με το λογιστικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκινάμε από τον λογιστικό έλεγχο δηλαδή. Συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια συστηματική επαλήθευση των αρχών λογιστικού ελέγχου στα κράτη-μέλη. Για το θέμα τώρα των κοινών κανόνων Θελήσαμε κοινού κανόνες για τα πέντε ταμεία. Μερικές φορές είναι κοινοί με πολλές λεπτομέρειες. Το θέμα της επιλεξιμότητας, για παράδειγμα, είναι ο ίδιος κανόνας που ισχύει για τα πέντε ταμεία με πολλές λεπτομέρειες και υπάρχει και απλοποίηση όσον αφορά το κόστος. Τώρα για το θέμα της διαχείρισης και του ελέγχου υπάρχουν κοινοί κανόνες σε επίπεδο αρχών, αλλά όχι πάντα και σε επίπεδο λεπτομερούς εφαρμογής. Γιατί πρέπει να υπάρχει και σταθερότητα των μηχανισμών. Και αυτό έχει να κάνει με την ε, ύπεθρο πρώτα απ' όλα, ανάπτυξη της ύπεθρου και πρέπει να διατηρηθεί. Πάντως για τα δύο σημεία τα οποία αναφέρθηκαν όσον αφορά την εκαθάριση λογαριασμών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, ότι η διαδικασία αυτή καθάρισης λογαριασμών θα συνεχίσει να θυχραμίζεται με τους στόχους, δηλαδή ότι οι λογαριασμοί είναι σωστοί, αλλά και ότι οι διάφορες συναλλαγές είναι κανονικές και νόμιμες, και αυτό σε διάφορους τομείς πολιτικής. Όσον αφορά τώρα τις δημοσιονομικές διορθώσεις, παρόλο που υπάρχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά τις λεπτομέρειες, τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να έχουν τα δικαιώματά τους και εγγυώνται ότι τα επίπεδα διόρθωσης ανταποκρίνονται και αντιστοιχούν με τα επίπεδα λάθους που έχουν τοπιστεί. Τώρα, απλοποίηση. Αυτή είναι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήθελε να επικεντρωθεί από την αρχή στην απλοποίηση για τους δικαιούχους, γιατί οι δικαιούχοι δεν πρέπει να τιμωρούνται όταν ζητούν χρηματοδότηση. Είχαμε όμως στο μυαλό μας επίσης και την μείωση του βάρους για τα κράτη-μέλη. Για να απαντήσω στον κύριο Ντί, έχουμε επιτελέσει μελέτη για, τα για το διοικητικό κόστος στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Τα αποτελέσματα θα τα έχουμε σύντομα και ευχαρίστως να σας θα δώσουμε στην Επιτροπή σας. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει κάποια βήματα μπροστά όσον αφορά την ε, απλοποίηση. Αναφέρθηκε το θέμα της ηλεκτρονικής η e-cohesion. Είμαστε όμως και ε, ανοιχτοί να συνεργαστούμε με τους συνομοθέτες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για να πάμε ακόμα πιο μακριά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα το ελεκτικό συνέδριο να αντιδράσει. Ίγκεμπορτ, έχεις κάτι να πεις? Ε, θέλω να πω κάτι στον κύριο Μάρτιν. Κοιτάξτε, αυτό που εντυπωσιάζει ε, και το αναφέρει επανειλημμένα το ελεγκτικό συνέδριο στη γνωμοδότησή του είναι το εξή. Ε, οι εξηγήσει ε, και το υλικό που ζητάμε, η δήλωση αξιοπιστία, αυτά πρέπει να είναι καλά συντονισμένα μεταξύ του. Γιατί υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Ποια είναι αυτή η δήλωση και ποιος θα κάνει εκ των υστέρων τι. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα γιατί αλλιώς ε, δεν θα είναι καλά τα χαρτιά μας όταν ζητάμε από τα κράτη-μέλη αυτές τις δηλώσεις αξιοπιστίας. Ε, θα πρέπει όλα αυτά να έχουν νόημα και τα στοιχεία να είναι αξιόπιστα. Αυτά έχω να πω αυτή τη στιγμή, αλλά αυτά που λέω δεν τα βλέπω να υπάρχουν στο σχέδιο που έχει κατατεθεί. Φαντάζομαι ότι σας άκουσε ο εισηγητής. Τώρα το ελεκτικό συνέδριο έχει την ευκαιρία να αντιδράσει. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή για να κλείσει, ποιος θα ξεκινήσει, ο κύριος Κρατένο ή ο κύριος Φαζάκας. Ποιος. Ο παλιός πρόεδρος της Επιτροπής μας, ε, ο κύριος Φαζάκας, που τώρα βέβαια είναι μέλος του ελεκτικού συνεδρίου. Έχετε το λόγο, παρακαλώ κύριε Φαζάκα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, ευχαριστώ που μου θυμήσατε την παλιά μου ιδιότητα ε, και με αυτή μου την ιδιότητα ερωτώ πόσο χρόνο έχουμε να εξτάσουμε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί, εντάξει, εγώ ε, να τοποθετηθώ, αλλά ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή γι' αυτό θα είμαι και πολύ σύντομο. Ε, πρώτον, σε ευχαριστώ πολύ για τι παρατηρήσει όσον αφορά τη γνωμοδότηση. Δεύτερον, όπω είπα και στην αρχή, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν είναι μόνο ευρύ, είναι και πολύ σημαντικό το θέμα που μπορεί να καθορίσει και το μέλλον της Ευρώπης από το 2014 μέχρι το 2020. Ε, κατόπιν τούτου, επιτρέψτε μου να πω και πάλι ότι εσείς λαμβάνετε αποφάσεις, εσείς είσαστε οι πολιτικοί, ε, εμείς ε, ως ελεγκτικό συνέδριο προσπαθούμε να σας διακονούμε, ε, να υποβάλουμε τις προτάσεις μας ε, και να ελπίζουμε ότι θα τις λάβετε υπόψη σας. Ο τελικός νομοθέτης που είστε εσείς ε, φαντάζομαι ότι ε, τα λαμβάνετε όλα αυτά ε, σοβαρά υπόψη. Αυτά γενικά. Και γι' αυτό το λόγο, όπως είπε πολύ σωστά και ο συγητή σας, ε, αποφάσισα, απέφυγα να πω ότι η μακροοικονομική αιρεσιμότητα είναι μεγάλο λάθος. Εμείς ε, ως ελεγκτικό συνέδριο το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν είναι ο σωστός τρόπος ε, ε, λύσης προβλημάτων. Δηλαδή όταν ένα κράτος αντιμετωπίζει μακροοικονομικά προβλήματα, το θέμα δεν είναι να του στερήσουμε κονδύλια από τα ταμεία. Εμείς ως ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να υπογραμμίσουμε πόσο σημαντικό είναι να μην συγχέονται δύο επίπεδα ελέγχου. Και εσείς, ε, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Γκρέσλε, και εμείς ε, καλούμετα να αναστείλουμε ε, πληρωμές αν ο δικαιούχος ε, κάνει, προβεί σε μία παρατυπία. Αυτό όμως είναι θέμα δικαιούχο. Όμως το να το αφαιρέσουμε κονδύλια λόγω μακροοικονομικών συνθήκων αυτό προκαλεί πολλά νομικής φύσεως οικονομικά προβλήματα σε επίπεδο επενδύσεων. Γι' αυτό λοιπόν με χαρά μας διαπιστώνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σέβεται όλα αυτά. Όσον αφορά αυτά που είπε η κυρία Γκρέσλε ε, σχετικά με το συντονισμό στο Ταμείο, αυτό το θέλουμε και εμείς. Και ε, και εμείς με μεγάλη μας απογοήτευση ακούσαμε ότι ο κανονισμός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ε, τα ταμεία με διαφορετικό τρόπο. Κατανοούμε τη θέση της Επιτροπής και επιθυμούμε να ευχηθούμε καλή τύχη στο Συμβούλιο έτσι ώστε ε, τα ταμεία τα οποία μοιάζουν τόσο πολύ να εναρμονιστούν μεταξύ τους ε, και έτσι ώστε ε, μια χώρα να μπορεί να υποφεληθεί. Τέλος, να σας πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς με όλα αυτά που ελέγχθησαν συμπεριλαμβανομένου και τον παρτιζόν κ. Μάρτιν ο οποίος μας εξήγησε πόσο πολύ ενδιαφέρεται στο να εφαρμόσει τις ε, συστάσεις του Συνεδρίου και του Κοινοβουλίου γιατί είχαν την καλοσύνη να μας καλέσουν στις ε, εργασίες ε, προετοιμασίες. Εμείς με μεγάλη μας χαρά ακούμε πάντα τις παρατηρήσεις του Συνεδρίου και του Κοινοβουλίου. Εσείς είστε οι νομοθέτες. Γι' αυτό λοιπόν όλοι μας ας ε, σκεφτούμε, ας, ας έχουμε κάποιο καλύτερο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, ο εισηγητής ε, θέλει να λάβει το λόγο γιατί έχουμε ήδη μισή ώρα καθυστέρηση και στις 12.30 πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Παρακαλώ. Ναι, θα είμαι πολύ σύντομο. Θέλω να απαντήσω στην κυρία Γκρέσλερ. Συμφωνώ με τα όσα είπε για την διαπίστευση και με τον κύριο για την απλοποίηση. Για το θέμα της επιμερισμένης ευθύνης περιμένουμε τα αποτελέσματα, όπως ε, μας είπε και η κυρία Γκρέσλερ. Τώρα όσον αφορά όσα είπε η Επιτροπή για το θέμα του κάπινγκ, τον, ανώ, τον καθορισμό ανωτά των ορίων δηλαδή. Θα έπρεπε να ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να είναι περισσότερο πρόβλημα για τις μεγάλες, ε, ε για τις μεγάλες χώρες, όσο για τις ε, μικρές Να δούμε λοιπόν τι θα προταθεί και ποιες θα είναι τελικά οι συνέπειες. Πάντως για τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα ε, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Δηλαδή έχει διαφορετική άποψη η Κομισιόν και διαφορετική άποψη έχουμε εμείς. Για το θέμα της διαπίστευσης είπα και στην αρχή ότι συμφωνώ επί της αρχής. Νομίζω ότι όντως είναι ε, κάτι καλό. Το βασικό είναι αν έχουμε διαπίστευση να ξέρουμε ότι την ευθύνη για τα κοινοτικά κονδύλια την τελική την έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία, λοιπόν, έχει επιτευχθεί πράγματι κάποια πρόοδος για τον επόμενο γύρο της ε, περιφερειακής πολιτικής, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν κάποια άλλη τα ζητήματα και ελπίζουμε στην επόμενη συνεδρίασή μας να έχει κάτι παραπάνω. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για όλο τον κόπο που έχετε κάνει για αυτό το θέμα. Οπότε έληξε έτσι το σημείο 12 στην ημερήσια διάταξη και τώρα περνάμε στο σημείο 13. 13 μέχρι 34, έτσι, είναι όλοι οι οργανισμοί. Η κυρία Μακοβέη είναι η συγγήτρια θα μας ε, το παρουσιάσει. Έχουμε και τον κύριο Σία, δεν απατώμε από το ελεγκτικό συνέδριο. Και θα δώσω και την ευκαιρία βέβαια και στους ευρωβουλευτές εδώ να παρέμβουν. Η Σιλβή για παράδειγμα. Αλλά και θα δώσω το λόγο και σε εκπροσώπους των ευρωπαϊκών αυτών οργανισμών που τους έχουμε εδώ. Κυρία Μακοβέη, έχετε το λόγο. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας έτσι, οπότε σας παρακαλώ κάποια πειθαρχία παρακαλώ. Η κυρία Μακοβέη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, καταρχήν όσον αφορά τους οργανισμούς. Διαπιστώνω ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού. Πήγαν από 3 στους 24 και σήμερα είναι 27 Ας δούμε λιγάκι ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία φτιάχνεται ένας ευρωπαϊκός οργανισμός. Γι' αυτό ευθύς εξ αρχής πρέπει να σας πω ότι πρέπει να το δει αυτό η Διοργανική Επιτροπή για την ε, δημιουργία νέων οργανισμών. Ελπίζω να καταλήξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε συμπεράσματα. Τώρα τι σημαίνει αυτό ε, περισσότεροι οργανισμοί σημαίνει και περισσότερα λεφτά. Έτσι. Το 2010 για τις 24 ε, τότε ευρωπαϊκές υπηρεσίες ήταν 1,5 δις περίπου ε, δισεκατομμύρια και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε με πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ. Τι βλέπουμε λοιπόν περισσότερους οργανισμούς ε, περισσότερα χρήματα. Αν χρειάζονται περισσότερα χρήματα πρέπει να δαπανώνται και υπεύθυνα. Είμαστε σε οικονομική κρίση, τα κράτη-μέλη υιοθετούν μέτρα λιτότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οργανισμοί πρέπει και αυτοί να είναι πολύ προσεκτικοί. Το συστήνω αυτό λοιπόν στο σχέδιο εκθεσή μου. Λέω δηλαδή ότι πρέπει να μην αυξάνονται άλλο οι ευρωπαϊκοί αυτοί οργανισμοί, να μην αυξάνεται άλλο ο προπολογισμό και μάλιστα να εξετάσουμε και τη δυνατότητα μείωση του προπολογισμού των ευρωπαϊκών αυτών οργανισμών, αξιολογώντα τι πραγματικέ ανάγκε των οργανισμών αυτών και ιδιαίτερα ε, όσον αφορά τους ερευνητικούς οργανισμούς. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει ένα κατάλογο προτεραιοτήτων για τις ανάγκες των ε, οργανισμών αυτών. Επίσης ζητάω από τους οργανισμούς να μειώσουν τα έξοδα λειτουργίας τους, να δουν ποια είναι ε, τα πραγματικά, τις πραγματικές τους ανάγκες και να εξετάσουν με λεπτομέρεια πού δαπανάτε κάθε ευρώ για τις μεταφορές, τα carry-overs. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλο ποσό εκεί, ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ακυρώσεις για το οικονομικό έτος 2010 από πολλούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Μπορώ να σας δώσω εδώ κάποια παραδείγματα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα Χημικά, για την Ασφαλή στη Θάλασσα, ε, η Ακαδημία Αστυνομίας. Και θα επαναλάβω εδώ αυτό που λέω και στην έκθεση, ότι λυπούμε που το λεκτικό συνέδριο δεν έχει αναφερθεί στην μεταφορά των πιστώσεων υποχρεώσεων που ακυρώθηκαν ή έχουν μεταφερθεί. Για τις δημόσιες προμήθειες επίσης και εκεί τίθεται θέμα για τις διαδικασίες. Ε, τώρα, σύγκρουση συμφερόντων. Κατά τη γνώμη μου, αλλά και για όλους μας, είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, μια που ορισμένοι συνεργάζονται με τη βιομηχανία. Το 2010 πολλοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί επικρίθηκαν στο σχέδιο έκθεσης ακριβώς επειδή υπήρξε σύγκρουση συμφερόντων. Ε, σημειώνουμε επίσης ότι το άρθρο 16 του υπηρεσιακού ε, κανονισμού δεν εφαρμόζεται πάντα. Υπάρχουν παραδείγματα σύγκρουση συμφερόντων πολύ συγκεκριμένα που θα τα βρείτε στα σχέδια ε, έκθεσης που υπάρχουν ε, για την υπηρεσία τροφίμων, φαρμάκων και περιβάλλοντος. Ε, για τον εσωτερικό έλεγχο τώρα. Θα ήθελα Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ καλή συνεργασία και να εκφράσω και την άποψή μου επ' αυτού. Όσον αφορά την Υπηρεσία εσωτερικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή η Επιτροπή βοηθάει τους οργανισμούς. Δηλαδή, αν διαπιστώσουν κάποιο πρόβλημα, ε, έρχονται σε επαφή με τον οργανισμό, όχι δημόσια βέβαια, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ως εκ τούτου, οι εκθέσεις ε, του εσωτερικού ελέγχου δεν δημοσιεύονται. Τώρα, αν δούμε λιγάκι το ε, πώς αντιμετωπίζονται οι εκθέσεις. Ε, οι εκθέσεις αυτές ε, λαμβάνονται υπόψη από τους οργανισμούς μόνο εφόσον το επιθυμούν οι διευθυντές και το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλιώς δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη. Βεβαίως μπορεί να υπάρξει γνωμοδότηση από το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι ένα λάθος στον κανονισμό που πρέπει να διορθωθεί. Κατόπιν, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, διαπίστωσα ότι υπάρχουν ε, δυστυχώς ε, πολλά διοικητικά συμβούλια με πολλά μέλη και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματικότητα. Εγώ δεν είμαι πεπισμένη ότι όλοι αυτοί είναι απαραίτητοι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός τους και επίσης και οι συνεδριάσεις τους είναι δαπανηρές. Τώρα, όσον αφορά τις πηγές πληροφοριών ε, που χρησιμοποιήθηκαν ε, σε αυτή την έκθεση και στην έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου, και εκεί ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Γνωρίζοντας βέβαια ότι το ελληνικό Συνέδριο έχει εκφράσει έχει ε, επικρίνει, έχει ασκήσει κριτική στη δική μου την έκθεση. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο είναι ο εξωτερικός ε, οργανισμός ελέγχου των οργανισμών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η υπηρεσία που δίνει την απαλλαγή. Χρησιμοποιούμε το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά για μας δεν είναι η μόνη πηγή ενημέρωσης. Κατόπιν του πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω χρησιμοποιήσει και πολλές άλλες πηγές ε, ενημέρωσης και όχι μόνο τις εκθέσεις του ελεγκτικού συνέδριου. Παραδείγματα, πρόγραμμα εργασίας, πρόγραμμα, ετήσιο πρόγραμμα δράση. προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωσης ε, του 2010, εκθέσει ε, από εσωτερικού ελεγκτές, ε, ίντερνετ και άλλε πηγέ πληροφόρηση. Και θέλω να σα πω ότι εφέτο, δυστυχώ, η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ήταν πολύ φτωχή σε επίπεδο ενημέρωση. Παραδείγματο χάρη για το 2010 το συνέδριο έδωσε μόνο 38 σχόλια ενώ το 9 69 σχόλια για 22 οργανισμούς. Παρότι λοιπόν υπήρχαν περισσότεροι οργανισμοί, τα σχόλια περιορίστηκαν ε, κατά το ίμιση. Επίσης, ε, το, τα σχόλια του ελεγκτικού συνεδρίου ε, περιλαμβάνουν έτσι γενικές τοποθετήσεις και όχι συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και θα ήθελα εδώ να κάνω και το εξής σχόλιο το ελεγκτικό συνέδριο, επειδή είναι ο εξωτερικός ελεγκτής, οφείλει να ενημερώνει ε, την κοινή γνώμη πρέπει να δίδονται πληροφορίες ε, ε, προς τα έξω και βεβαίως και στην αρχή απαλλαγής, χωρίς απαλλαγής. Τώρα μερικά για την έκθεση για το benchmarking. Στο ελεγκτικό συνέδριο σχεδιάζεται να δημοσιευτεί χωριστή έκθεση για αυτό το θέμα το 11. Είχε προβλεφθεί. Δεν την είδαμε όμως αυτή την έκθεση. Τη ζητήσαμε πολλές φορές. Δύο εβδομάδες πριν λάβαμε μία επιστολή προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου με την οποία επισυναπτόταν ένα έγγραφο που έλεγε ότι δεν πρόκειται για την έκθεση benchmarking, δεν είναι δημόσιο έγγραφο και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για, ως βάση εκθέσεων. Αυτό δεν μου φαίνεται σοβαρό, γιατί δεν έγινε η έκθεση benchmarking όπως προβλεπόταν το 2011. Πάρα, πήραμε μόνο μια επιστολή με μερικούς αριθμούς και που δεν έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε. Τώρα για μεμονωμένες εκθέσεις για τις υπηρεσίες και τα ιδρύματα δεν συμπεριέλαβα τις απαλλαγές τους στην έκθεσή μου γιατί ήθελα πρώτα να έχω περισσότερες πληροφορίες από τα Ιδρύματα και πρέπει να σας πω ότι συνάντησα εκπροσώπους πολλών εξ αυτών την το Ιατρικό Ίδρυμα, το Ίδρυμα, την Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων και άλλα. Και αύριο θα συναντήσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Νομίζω ότι είναι καλό να συνομιλούμε με τους διευθυντές των υπηρεσιών αυτών. Με μερικούς συνομίλησα από το τηλέφωνο και είναι καλό να έχουν τη δυνατότητα και αυτοί να σχολιάσουν το σχέδιο έκθεσης. Τις ευχαριστώ λοιπόν όσες συνεργάστηκαν. Θα σταματήσω εδώ για τις υπηρεσίες και τα ιδρύματα για να ακούσω για να ακούσω, για να ακούσω. Εσείς τώρα. Θέλετε να συνεχίσω. Αν θέλετε μπορείτε να συνεχίσετε για το επόμενο θέμα. Μπορείτε, ίσως είναι προτιμότερο, πιο εύκολο όλα μαζί να τα δείτε. Ωραία, το επόμενο είναι η απαλλαγή για το 2010 των κοινών επιχειρήσεων δεν είναι κάτι με το οποίο είμαστε πολύ εξοικειωμένοι. Δίνουμε απαλλαγή στις κοινέ επιχειρήσεις. Νομίζω ότι τα όλα στους φακέλους σας με τις 7 κοινέ ε, επιχειρήσεις που έφτιαξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρούν σε έρευνες σε διάφορους τομείς. Έξι από τις 7 ε, κάνουν έρευνες και μία ασχολείται με τη διαχείριση του νέου συστήματος ε, αεροπορικών μεταφορών, τη G-Move. Είναι πολύ υψηλά τα ποσά. Οι πόροι που κρίνει αναγκαίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 10 χρόνια είναι οι με κάποιες εξαιρέσεις. Τα βλέπετε στους πίνακες, οπότε η συνολική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Και για το οικονομικό έτος 2010 η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον προπολογισμό τους ήταν πάνω από 500 εκατομμύρια για ένα έτος δηλαδή. Υπάρχουν εταιρικέ ε, σχέσεις δημοσίου και ιδιωτικού ε, τομέα οργανώσεων δηλαδή, οπότε παίρνουν χρήματα και από τον ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά τώρα την ενημέρωσή μας. Έχω από το ελεκτικό συνέδριο, από την εκθεσή του δηλαδή, που πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την περίπτωση μας έδωσε πάρα πολλές πληροφορίες. Βρίσκω δηλαδή ότι είναι πολύ καλή η εκθέση αυτή και πλήρης. Πήρα πληροφορίες επίσης και από την προσωρινή αξιολόγηση των ετησίων δραστηριοτήτων των κοινών ε, αυτών επιχειρήσεων, αλλά και από επαφές που είχα. Η απόφαση για την ε, απαλλαγή θα αποφασιστεί μέσω των τροπολογιών, βασιζόμενοι βέβαια και στις αντιδράσεις που θα έχουμε στο σχέδιο έκθεσης. Στην, στην κάθε έκθεση για τις ε, μικτές επιχειρήσεις θα δείτε ότι υπάρχει ένα οριζόντιο τμήμα, το τελευταίο τμήμα, το οποίο είναι κοινό και για τις 7. Ελπίζω του χρόνου να υπάρξει μια οριζόντια έκθεση για τις επιχειρήσεις αυτές. Υπογραμμίζω επίσης αυτό το οριζόντιο τμήμα τις ελλείψεις που διαπίστωσα σε όλες τις κοινέ επιχειρήσεις και αυτό έχει να κάνει ότι είναι πολύ ψηλό το επίπεδο των μεταφορών, το κέρι offense, όπως επίσης και του ρευστού, οι ακυρώσεις αναβολές των υποχρώσεων, η τήρηση αρχών μερικές φορές για τις προμήθειες και σχετικά με τις πληρωμές που γίνονται από τα κράτη-μέλη. Συνεπώς, και εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για τη σύγκρουση συμφερόντων. Οι επιχειρήσεις αυτές είπαμε ότι είναι συνδυασμό ιδιωτικού δημοσίου. Άρα ε, τα συμφέροντα εδώ κάπου συναντιόνται. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε διάλογο με τις εκείνες αυτές επιχειρήσεις, ακόμα και αν ε, είμαστε επικριτικοί. Το ίδιο ισχύει και για το ελεκτικό συνέδριο. Ε. Και θα ήθελα να ακούσω τώρα τους διάφορους οργανισμούς αλλά και τους συναδέρφους και να ολοκληρώσω λέγοντας, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν επικρίσεις, να πω λοιπόν ότι η κριτική μας βοηθάει να προχωράμε περισσότερο. Όποιος θέλει, υποβάλλει τροπολογίες και μετά θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μακοβέη. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σύ από το Ελεγκτικό Συνέδριο πρώτα απ' όλα. Από ό,τι κατάλαβα είναι η προτελευταία σας μέρα στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Κάνατε τον κόπο να έρθετε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ και κυρίως σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη δουλειά που έχετε κάνει. Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά μαζί, πολύ καλές σχέσεις έχουμε τα θα δώσω βέβαια στην εισηγήτρια. Τώρα πολλές ερωτήσεις τη εισηγήτρια. Σίγουρα θα έχετε και εσείς πολύ καλές απαντήσεις. Σας ακούμε. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Στάση. Ευχαριστώ την κυρία Μακοβέη για τη συνεργασία μας καθ' όλη την περίοδο που εκείνη ήταν η και εγώ αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά ιδρύματα. Είναι μεγάλη τιμή η παρουσία μου σήμερα εδώ για την παρουσίαση 29 δημοσίων εκθέσεων του συνεδρίου φέτος. Οι εκθέσεις αυτές είναι δημόσιες, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας και στην επίσημη εφημερίδα. Επίσης, ευχαριστώ τον κύριο Στάις που θέλησε να συζητήσουμε το θέμα της έκθεσης benchmarking, η οποία υποβλήθηκε πριν από δύο εβδομάδες. Αν έχετε απορίες παρακαλώ να μου τις πείτε. Αν έχετε πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να σας είναι χρήσιμες, θα ήθελα να σας πω ότι ξέρουμε ότι το Κοινοβούλιο συχνά έχει ζητήσει πληροφόρηση για τις υπηρεσίες και τα Ιδρύματα και πάντοτε τις χορηγούσαμε. Μάλιστα δημοσιεύσαμε περισσότερες πληροφορίες φέτος για τις υπηρεσίες από ό,τι πέρυσι. Παρά το ότι εγώ μόνο δύο χρόνια ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Υπήρξε παρόλα αυτά σημαντική αύξηση. Αυτό είναι γεγονός. Εκτός από τις εκθέσεις που δώσαμε, γίνανε και επαφές μεταξύ ελεγκτικού συνεδρίου και των αρχών που είναι αρμόδιες για τον προϋπολογισμό ως προς την απαλλαγή των υπηρεσιών. Επιστολές προς τον Πρόεδρο και του Προέδρου σε απάντηση ερωτημάτων το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο και στις 16 Φεβρουαρίου φέτος. για να δούμε πώς τα πήγαν γενικά οι υπηρεσίες και τα ιδρύματα φέτος, εμείς παρατηρήσαμε μία βελτίωση στην αποτελεσματικότητά τους. Ιδιαίτερα τονίζω το θέμα του Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, που επί πολλά χρόνια ήταν προβληματική αλλά είχα ακούσει και την πρώτη φορά που ανέλαβα το θέμα την κυρία Μάθιου να αναφέρει τα προβλήματα και πέρυσι ο ίδιος μίλησα δημόσια πολύ επικριτικά για την αποτελεσματικότητά της το 2009 αλλά φέτος πρέπει να σας πω ότι τα πράγματα σημαντικά βελτιώθηκαν Εμείς τώρα στο συνέδριο θεωρούμε την υπηρεσία αυτή σαν μία από τις υπηρεσίες με το χαμηλότερο κίνδυνο, πράγμα που δεν συνέβαινε πριν από δύο και τρία χρόνια πριν και τα προηγούμενα όσες φορές επικρίναμε τους, τη διαχείρισή της. Η Ευρωπαϊκή Ιατρική Υπηρεσία και πέρυσι και φέτος δεν σημείωσε κανένα προβλήμα. Έκανε πολλή δουλειά για τα δημοσιονομικά της και αυτό είναι βελτίωση επίσης σε σύγκριση με πέρυσι. Γενικά υπήρξε βελτίωση στην αποτελεσματικότητα και λειτουργία και διαχείριση των υπηρεσιών. Τα ίδια προβλήματα σημειώνονται κάθε χρόνο. Οι προμήθειες, οι προσλήψεις. Καιρός είναι οι υπηρεσίες να τα λύσουν αυτά τα προβλήματα και πιστεύω ότι το έχουν προσπαθήσει μαζί με το Κοινοβούλιο και τις επικρίσεις του και με τις επικρίσεις του συνεδρίου για να λύσουν τα προβλήματα που απομένουν και που δικαιολογούν τις συχνές αυτές επικρίσεις. Είναι καλό ότι τα αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα γιατί αυτό αναμένει και το κοινό να λύνουν τα προβλήματα. Το συνέδριο έχει συγκεκριμένη εντολή να δηλώνει ό,τι βλέπει άφοβα. Αυτό ακριβώς κάνουμε επαγγελματικά σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και με τις ευθύνες που μας έχουν ανατεθεί από τις συνθήκες. Δημοσιεύσαμε μια έκθεση με τίτλο Cost Benchmarking. Η κυρία Μακοβέη μας είπε ότι θελήσαμε να παραμείνει εμπιστευτικό, εμπιστευτική έκθεση. Αυτή παρόλα αυτά διέφυγαν πολλά στα μέσα ενημέρωσης. Από την έκθεση αυτή δόθηκε η εντύπωση ότι 11 από τις 22 εποπτικές αρχές δεν δικαιολόγησαν σωστά τις δαπάνες τους. Εγώ νομίζω ότι αν διαβάσετε καλά την έκθεση αυτή θα δείτε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και με την ευκαιρία αυτή πρέπει να σας πω σήμερα ότι η λογοδοσία των υπηρεσιών βασίζεται στους λογαριασμούς τους. Και οι 22 έλεγχοι το 10 κατέληξαν σε αξιόπιστα στοιχεία και τους λογαριασμούς αυτούς δεν τους θεωρούμε λανθασμένους. Δεν μου αρέσει να λέγονται άδικα πράγματα και πρέπει να σας πω σήμερα ότι οι επόπτες, οι ελεγκτές δεν έχουν πει ποτέ τίποτα τέτοιο όπως αυτό που υποτίθεται ότι λέγαμε στην έκθεση benchmarking. Εδώ πρόκειται για λάθος ή παραπληροφόρηση. Κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι μπορώ να αποφύγω εδώ ορισμένα σχόλια για μερικά από αυτά που είπε η κυρία Μακοβέη στην έκθεσή της για τις υπηρεσίες. Ιδιαίτερα ως προς το ελεγκτικό συνέδριο. Υπήρξαν πολλές ανταλλαγές επιστολών μεταξύ Κοινοβουλίου και ημών και εμείς στο συνέδριο πάντοτε ασμένος δεχόμαστε τέτοιες επιστολές. Την περασμένη εβδομάδα στις 22 Φεβρουαρίου πήραμε την τελευταία και μάθαμε ότι το σχέδιο έκθεσης δεν είναι αναγκαστικά η άποψη της κοκομπούς. Γιατί όλοι και εμείς και εσείς εφαρμόζουμε ανεξάρτητα και επαγγελματικά κριτήρια και είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ συνεδρίου και επιτροπής σας. Είμαι εδώ και δύο χρόνια στο συνέδριο, είχαμε εξαιρετική συνεργασία για οποιοδήποτε θέμα τέθηκε. Γιατί όταν συνεργαζόμαστε ωφελούνται οι λαοί της Ευρώπης. Αν έχετε απορίες με τα χαράς να τις ακούσω και σας ευχαριστώ εκ νέου κύριε Πρόεδρε και κύριοι βουλευτέ για τη συνεργασία μας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και τόσο ευθύς. Τρεις έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Ματιέ, ε, η κυρία Χέτσοκ και ο κύριος Γκεμπραντή, ο οποίο βέβαια βγήκε λίγο γιατί στις παρατέταρτο έχει ένα ραντεβού με την τηλεόραση. Φαντάζομαι ότι θα γυρίσει πίσω. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυρία Ματιέ. Α, Διακόπτει ο πρόεδρος. Το ΕΛΚ πήρε το λόγο, όντως, οπότε θα το δώσω στους σοσιαλιστές τώρα. Κυρία Χέρτσοκ, εσείς, με αυτή τη σειρά. Ναι, κανένα πρόβλημα. Νόμιζα ότι πήγαινε με τη σειρά που ζήτησε κανείς το λόγο, αλλά τόσο πάντων δεν έχει σημασία. Δεν είναι πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς θέλω πολύ να ακούσω την άποψη της κυρίας Ματιέ. Θυμάμαι πριν από τρία χρόνια ήμουν εγώ εισηγήτρια για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και το θυμάμαι. Είναι αλήθεια ότι τώρα έχουμε περισσότερους ακόμα οργανισμούς. Βλέπω όμως επίσης ότι αυτά τα τρία χρόνια υπάρχει μεγάλη προστιθέμενη αξία στο έργο των οργανισμών αυτών. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Η συγγήτρια, μάλλον κάποιος εισηγητής που έχει αναλάβει μία φορά την έκθεση αυτή για τους οργανισμούς γνωρίζει πάρα πολύ καλά πόσο τεράστιο είναι το έργο αυτό. Ακριβώς επειδή έχουμε τόσους πολλούς οργανισμούς. Είναι δηλαδή μια ειδική έκθεση αυτή, ένα ειδικό θέμα. Πάρα πολλή δουλειά και πολλές θυσίες για να ετοιμαστεί η σύσταση αυτή. Η κυρία Μακοβέη λοιπόν πιστεύω ότι δούλεψε πολύ Και επίσης ίσως χρειαζόμαστε τα επόμενα χρόνια περισσότερο χρόνο προκειμένου και οι σκιώδες εισηγητές να ετοιμάζουν την άποψή του ακριβώς γιατί είναι πάρα πολλή δουλειά. Καταλαβαίνετε ότι αν οι σκιώδες πρέπει να ετοιμάσουν τη δικιά τους την τοποθέτηση, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχουμε το χρόνο για να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, είναι περισσότεροι μεν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, πιο ορατοί, προβάλλονται περισσότερο στους πολίτες. Είναι όμως το 47%. Ακόμα και οι μικροί και οι μεγάλοι έχουν μεγάλες επιπτώσεις όσον αφορά τις πολιτικές μας. Ιδιαίτερα οι οι κοινέ επιχειρήσεις. Οι κάνουν έρευνα και το θυμάμαι από την Επιτροπή Βιομηχανία που λέμε ότι φέρουν σε πέρα τους στόχους τους, έχουν αποτελέσματα και βελτιώνουν τις επιδόσεις των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάθε μία στο δικό της τον τομέα. Καλά, αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα, αλλά λέω ότι η Επιτροπή ότι αυτού του είδους οι οργανισμοί φέρνουν αποτελέσματα. Έτσι για να σχηματίσετε ε, την εικόνα. Σήμερα είναι λιγότερο από το 5% του κοινοτικού προπολογισμού, οπότε πρέπει να δούμε τα πράγματα στην κανονική τους διάσταση. Όπως είπα, σε σύγκριση με το τι γινόταν πριν από τρία χρόνια που ήμουν εγώ εισηγήτρια, εξακολουθώ να σκέφτομαι και εγώ το ίδιο, ότι υπάρχει βελτίωση όσον αφορά τα αποτελέσματα. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Είναι πολλή δουλειά. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές από τότε που δημιουργήθηκαν οι οργανισμοί και στους περισσότερους έχουμε πετύχει αυτό που θέλαμε. Οι οργανισμοί που έχουν καλά αποτελέσματα πρέπει να εξάγουν εντό αγωγικών την ε, γνώση τους, τις ε, ικανότητές τους, έτσι ώστε να βοηθηθούν και άλλοι οργανισμοί. Γι' αυτό λοιπόν και αναρωτιέμαι με την επιστολή μου του Νευρίου προς το λεκτικό συνέδριο, μήπως θα έπρεπε να επικεντρωθούμε όχι μόνο στις αδυναμίες αλλά και στα θετικά των οργανισμών αυτών και να υπάρχουν και τα δύο δηλαδή στην έκθεση. Γιατί είναι θεμέλια πάνω στα οποία μπορούμε να χτίσουμε. Θέλω να μου απάντησε βέβαια το Δεκέμβριο ο κ. Καλτέρο πρόεδρος και αυτό βοήθησε πολύ και την Επιτροπή μας. Θέλω να επαναλάβω και κάτι άλλο για το ΣΥΠΟΛ. Και η ίδια κατάσταση ήταν για χρόνια. Ακριβώς επειδή είχαμε επειδή φροντίσαμε εμεί η Επιτροπή μας και η συγκήτρια η κυρία Ματιέ και νωρίτερα ο κύριος Φέλκνερ και χάρη και στη δουλειά του νέου Ούγγρου Προέδρου και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, βλέπουμε μεγάλη βελτίωση. Άρα είναι καλό να είμαστε επικριτικοί, αλλά συγχρόνως και πρέπει να είμαστε θετικοί. Βλέπουμε ότι αυτό που έγινε στον οργανισμό αυτό είναι καλό. Κάτι άλλο να πω για τη ΣΕΠΟΛ και τη Europol. Αναρωτιέται στην έκθεσή της η κυρία Ματιέ για τη ΣΥΠΟΛ αλλά όχι για τη Europol. Ίσως οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές θα πρέπει να ασχοληθούν με το περιεχόμενο και με τα καθήκοντα των δύο αυτών οργανισμών. Γίνεται λοιπόν πολλή δουλειά, πολλά θετικά. Έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και αναφέρονται στην έκθεση της κυρίας Μακοβέη. εισαγάγει όμως και κάποιες επικριτικές παρατηρήσεις. Σε αυτές θα αναφερθώ λοιπόν, ακριβώς γιατί προσπαθούμε να πετύχουμε ένα συμβασμό. να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος με την έκθεση απαλλαγής μας να τα να ενημερώσουμε το κοινό. Ελπίζω ότι η συγγήτρια θα είναι ανοιχτή απέναντί μας και θα συνεργαστεί στενά με τους σκιώδες εισηγητές για να καταλήξουμε σε ένα τελικό κείμενο και να καταλήξουμε σε συμφωνία. Λοιπόν, για τις επικρίσεις. Πρώτα απ' όλα αυτές του ελεκτικού συνεδρίου. Ζητάω από την εισηγήτρια λοιπόν οι επιστολές που έχουν ανταλλάξει είναι ικανοποιητικέ για εκείνη. Έπειτα, αν έχουμε μια γνωμοδότηση για τους άλλους οργανισμούς. Μήπως τις παρατηρήσεις πρέπει να τις βάλουμε στην απαλλαγή ε, της έκθεσης που κάνουμε για τον κάθε οργανισμό. Ένας από αυτούς είναι το ελεγκτικό συνέδριο. Ίσως πρέπει να σκεφτούμε είναι το καλύτερα σελίδα των οργανισμών ή τις παρατηρήσεις αυτές να τις βάλουμε στην έκθεση για τους άλλους οργανισμούς. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό κάποια στιγμή. Λυπάμαι που οι εισηγητές για τους άλλους οργανισμούς δεν είναι εδώ. Πέραν αυτού πάντως, υποθέτω ότι γενικά Μπορούμε να είμαστε γενικοί όταν μιλάμε για θετικά πράγματα, αλλά όταν έχουμε να πούμε κάτι αρνητικό πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Βλέπετε τα αρνητικά δεν κάνουν καλό όταν διατυπώνονται έτσι γενικά. Αν κάποιος έχει κάποια κριτική, να το πει συγκεκριμένα. Εγώ ε, είμαι γενική όταν έχω να πω κάτι θετικό, αλλά όταν βλέπω κάτι στραβό, το λέω πολύ συγκεκριμένα. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη προσέγγιση. Να είμαστε συγκεκριμένοι κάθε φορά που έχουμε μια επικριτική παρατήρηση και να μην γενικεύουμε. Προς αυτή την κατεύθυνση θα υποβάλω και εγώ κάποιες τροπολογίες για να βελτιώσω την έκθεση. Τώρα, συμφωνώ με την εισηγήτρια με τη γενική της προσέγγιση που λέει ότι ιδιαίτερα τώρα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε οικονομική κρίση πρέπει να γίνουν οικονομίες. Βεβαίως. Βεβαίως οικονομίες. Αλλά οικονομίες για το μέλλον είναι σε άλλη έκθεση. Έχουμε τον κανονισμό προσωπικού με την κυρία Κρέσλερ. Άρα να προσέξουμε πολύ ε, πόσο πολύ σε βάθος θα πάμε με τέτοιες παρατηρήσεις για τις εκθέσεις για τους οργανισμούς. Τώρα, οι μεταφορές, τα carry-overs, πρέπει να τα ξαναδούμε. Να ε, βελτιωθούν βέβαια, αλλά βλέπετε οι λόγοι είναι διαφορετικοί ανάλογα με τους οργανισμούς. Γιατί δηλαδή συμβαίνουν αυτές οι πολλές μεταφορές. Σίγουρα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Πάντως, οποιοδήποτε είναι τα ταμείας όπως είμαι εγώ στους σοσιαλιστές, και εγώ έχω πρόβλημα με τις μεταφορές αυτές. Είτε πρόκειται για τις αντιπροσωπείες, είτε για την ομάδα. Είναι κάτι που δεν αρέσει καθόλου στους ταμείες. Αλλά γι' αυτό ακριβώς καταλαβαίνω ότι οι αιτίε μπορεί να είναι εντελώ διαφορετικές. Γι' αυτό και λέω πάλι, όχι γενικότητες. Δεν θα μας βοηθήσουν. Αναφέρθηκε στη σύγκρουση εφερόντων επίσης η κυρία Μακοβέη. Πράγματι, είναι ένα πρόβλημα για τις κοινέ επιχειρήσεις και για τους πολιτικούς οργανισμούς. Όσο πιο ειδικευμένος είναι ο οργανισμός, τόσο πιο πολύ εμφανίζεται το πρόβλημα αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οποιοςδήποτε μπορεί να εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένας και ικανότητες για δουλειά. Είναι φυσιολογικό για κάτι όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά όταν μιλάμε για συγκεκριμένους οργανισμούς, για τα χημικά, για παράδειγμα, για το περιβάλλον, που και αυτά ακόμα ίσως γενικά, αλλά για τα φάρμακα ή την αεροπορία. Το πρόβλημα είναι ότι από τη μια μεριά θέλεις τους καλύτερους και από την άλλη μεριά δεν έχεις και τεράστια επιλογή. Αναπόφευκτα λοιπόν θα βρεις ανθρώπους που έρχονται από κάποιους σχετικούς τομείς. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο να επιλέξεις τον συγκεκριμένο και να δεις που θα δουλέψει, αλλά πρέπει να έχουμε και ένα πλαίσιο, διότι η δουλειά γίνεται συνήθως ομαδικά. Η ομάδα λοιπόν πρέπει να βρίσκει τη λύση, άρα δεν πρόκειται μόνο για το άτομο, πρέπει δηλαδή η οργάνωση να είναι τέτοια που να δουλεύουν μέσα σε ομάδα, οπότε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Θα ήθελα να το βάλω και αυτό ο οργανισμός. Τέλος, η συγγήτρια, αλλά... Θέλω να μιλήσω για τις συγχωνεύσεις. Η συγχώνευση σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι μια πολύ καλή ιδέα, οικονομικά, δημοσιονομικά. Αλλά μετά, αν κοιτάξουμε τους λόγους για τους οποίους δημιούργηθηκε ο κάθε οργανισμός είναι πολύ δύσκολο να έχουμε συγχώνευση. Γι' αυτό εδώ προτείνω να κάνουμε μία αξιολόγηση και αντί να αποφασίσουμε εμείς από μόνοι μας να το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τους διάφορους οργανισμούς και την Επιτροπή και τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές που ίδρυσαν τους οργανισμούς αυτούς ή τις μεικτές επιχειρήσεις και να το δούμε μαζί τους. Μάλιστα στην έκθεση για τις κοινέ επιχειρήσεις θα έλεγα να ζητήσουμε από τους ηχητές του ορίζοντα 2020 πώς το βλέπουν και πώς μπορούν να βελτιώσουν το έργο των διάφορων οργανισμών και των κοινών επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα θέματα τους. Αλλά να μην καταργήσουμε κάτι που θα έχει τελικά αρνητικές συνέπειες. Αυτές είναι οι σύντομες παρατηρήσεις μου και ελπίζω ότι θα βρούμε έναν τρόπο να συμφωνήσουμε και ελπίζω η κυρία Μακοβέη να είναι ανοιχτή για συνεργασία μαζί μας. Επαναλαμβάνω ότι οι σκιώδες εισηγητές θα πρέπει να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους. Και περισσότερη συνεργασία θα έλεγα στα αρχικά στάδια. Είπαμε, είναι ένα τεχνικό θέμα αυτό με πολλές ιδιαιτερότητες. Σε πολλές περιπτώσεις η διατύπωση ήταν διαφορετική σε αυτά που κάναμε εμείς από εκείνη που χρησιμοποίησε και η ορολογία που χρησιμοποίησαν οι δημοσιονομικές αρχές. Ή τα νομικά κείμενα διαφέρουν από τη δικιά μας την έκθεση στην ορολογία. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι για αυτές τις εκθέσεις όντως 6 Μαρτίου που είναι 5 Μαρτίου μάλλον είναι η προθεσμία έτσι ε, η ψηφοφορία θα γίνει μετά ε, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Ε, τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε λιγάκι. Αλλά εδώ αδίκησα λίγο το λεκτικό συνέδριο, γιατί μίλησε η κυρία Μακοβέ και για τις ε, κοινέ επιχειρήσεις. Ο κύριος Βάλκο είναι εδώ από το λεκτικό συνέδριο για αυτό το θέμα. Θέλετε να πάρετε το λόγο παρακαλώ. Αλλά βέβαια με πειθαρχία έτσι γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι υπεύθυνο για τις μικτές επιχειρήσεις και όπως ξέρετε αυτά τα joint undertakings είναι κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και όπως είπε και η κυρία Μακοβέη πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους όπως νέες οντότητες που πρωτοδημιουργήθηκαν το 2008 και με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και υψηλό προϋπολογισμό. παρά τις αρχικές τους δυσκολίες, μερικές από αυτές τις joint undertakings άρχισαν να λειτουργούν. Για το 10, που είναι και η βάση της έκθεσης μας σήμερα, τονίζω δύο πτυχές. Πρώτον, συμφωνούμε γενικά με, τις, με τα σχόλια του συνεδρίου για τα joint undertakings. Δεύτερον, τα σχόλια του συνεδρίου υποστηρίζονται και από το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Μακοβέη. Χαίρομαι για αυτή την επικοδομητική συνεργασία που θα ωφελήσει όχι μόνο τους δύο μας, τα δύο μας θεσμικά όργανα, αλλά και στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων. Επίσης χαίρομαι και ενθαρρύνομαι από την αναγνώριση της κυρίας Μακοβέη ότι τα σχόλια του συνεδρίου για το joint undertakings μας δίνουν χρήσιμες και επαρκείς πληροφορίες. Τέλος, δεν μπορώ να προσθέσω παρά μόνο ότι λάβαμε πλήρως υπόψη μας το αίτημα να κάνουμε ειδική έκθεση για τα joint undertakings. Η αποτελεσματικότητα ήταν το κριτήριό μας. Βέβαια το συνέδριο όλα αυτά τα αιτήματα τα λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του για να δει πώς μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα και ιδίως με τι χρονοδιάγραμμα και με τι μορφή. Σε ενιαία έκθεση, χωριστή ή όχι. Βέβαια πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη μας και το σχεδιασμό των εργασιών του συνεδρίου. Ο κύριος Φάζακας είναι ο υπεύθυνος και εγώ είμαι υπεύθυνος για την εποπτεία 6 μόνο joint undertaking. Σε ευχαριστώ. Κυρία Ματιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν συγχαίρω την κυρία Μακοβέη για τη δουλειά της Ξέρω ότι το θέμα της είναι κάτι που σημαδεύει οποιαδήποτε κοινοβουλευτική θητεία. Είναι τελείως ιδιαίτερο. Θα ήθελα να πω ότι οι υπηρεσίες αυτές και οι κοινέ επιχειρήσεις joint undertakings είναι κάτι πολύ χρήσιμο στην Ένωση. Δεν υποτιμώ καθόλου τη σημασία του προϋπολογισμού τους γιατί είναι πολύ χρήσιμες και για μας αλλά και για τους πολίτες της Ευρώπης. Αν η κυρία Μακοβέη προτείνει κριτήρια για τη δημιουργία και νέων, δεν θα ήμουν κατά αν και δεν θέλω να υπάρχουν υπερβολικά πολλές για να μην υπάρχει κατακαιρματισμός. Επίσης θα ήθελα να πω ότι η έκθεσή της λέει πολλά θετικά ιδιαίτερα όμως για το σε πόλ θέλω να ενδιαφερθώ και να καταθέσω τροπολογίες καθώς και για την υπηρεσία φαρμάκων και περιβάλλοντος ε, καθώς και μερικών τροφίμων. Να θα καταθέσω όμως σχετικά το πολύ, θα συνεννοηθώ με την κυρία Μακοβέη. Ήθελα επίσης να πω ότι οι διευθυντές των υπηρεσιών αυτών κάνουν κάτι πολύ χρήσιμο και πολλές φορές τα διοικητικά του συμβούλια δεν τους επιτρέπουν να δράσουν όπως θα ήθελαν Υπάρχει επίσης εδώ ένα θέμα διαμάχης αρμοδιοτήτων πράγμα το οποίο αναφέρει και η κυρία Μακοβέη σε μερικές υπηρεσίες όπως του περιβάλλοντος, των φαρμάκων και της τροφιμικής ασφαλείας. Θα ήθελα μερικές περισσότερες λεπτομέρειες επ' αυτού. Να, αυτά ήθελα να πω. Αλλά θέλω να μου απαντήσετε εδώ για το παντουφλάζι ιδίως, για το παντοφλάρισμα. Ευχαριστούμε κύριο Σκεμπραντή. Εντάξει με τηλεόραση, επιστρέψατε βλέπω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ναι. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση που δείχνετε. Θα αρχίσω με ευχαριστίες προς την κυρία Μακοβέη για τη δουλειά της. Όντως, είναι εντυπωσιακό ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά. Έχω βέβαια και διάφορα ερωτηματικά. Γιατί κατά τη γνώμη μου για αυτήν την κοινοβουλευτική επιτροπή αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να, είμαστε, να δουλεύουμε με ε, πολύ προσοχή αλλά και να είμαστε και απολύτως ανεξάρτητοι γιατί δεν ε, πρέπει να μπορεί κανείς ε, να μας ε, προσάψει τίποτα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ε, πολύ προσεκτικοί. Δεν ισχύει το ίδιο με όλες τις επιτροπές. Εμείς δεν είμαστε πολύ δημοφιλεί ε, απαραίτητα. Λοιπόν, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πώς δουλεύουμε. Εμείς δεν ε, είμαστε όπως το λεκτικό συνέδριο. Υπάρχει μια αν... ανεξαρτησία, αλλά εγώ δεν θέλω να πάω τόσο μακριά όπως ε, πάει και η κυρία Μακοβέ, η οποία αμφισβητεί, για παράδειγμα, την ανεξαρτησία του λεκτικού ε, συνεδρίου. έχει πολύ σημασία για το κύρος η δουλειά που κάνουμε. Δεν υπάρχει λόγος προς το παρόν κανένας να αμφισβητήσει τις προθέσεις μας ή τις προθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Η επιστολή εξάλλου του Πρόεδρου Καλντέρα είναι μια αντίδραση στην έκθεση Μακοβέη. Την έχω εδώ και βλέπω ότι τα διάφορα επικριτικά σημεία τα οποία πάνε πολύ μακριά πολιτικά θα έλεγα, ότι εκεί δίνει ο κύριος Καλντέρ εξηγήσει. Οπότε θέλω να ρωτήσω την κυρία Μακοβέη, θέλει να αντιδράσει σε αυτό ή είναι διατεθειμένη κάποια σημεία στην έκθεσή της να τα αποσύρει και κατά πόσο συμφωνεί με ε, την απάντηση του ελεγκτικού συνεδρίου. Το λεκτικό συνέδριο ε, λοιπόν, ήταν ένα σημείο. Τώρα, για την υπηρεσία περιβάλλοντος, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Και επιτίθεται στον οργανισμό αυτό, κυρία Μακοβέη, στην ε, έκθεσή της. Ομολογώ ότι με ξέπληξε. Εγώ έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Κοπεχάγη, την έδρα του οργανισμού αυτού και μου κάνει εντύπωση η καλή ποιότητα δουλειάς του οργανισμού αυτού. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του είναι κάτι το οποίο βρίσκω εγώ πραγματικά αξιοπρόσεχτο. Με εξέπληξε όπως σας είπα. Και ίσως η κυρία Μακοβέη εδώ ε, μπορεί να μου απαντήσει. Όπως επίσης και για την κριτική της που είναι σε όλη την ε, έκθεση. Το περιβάλλον είναι ένα παράδειγμα είναι ε, οργανισμός στον οποίο έχουμε πολλούς επιστήμονες. Οι επιστήμονες τι κάνουν, γράφουν εκθέσεις. Υπάρχουν ε, λοιπόν πολλά επικριτικά σημεία όσον ε, αφορά το, τον οργανισμό αυτόν περιβάλλοντος. Έχω και την απάντηση όμως του οργανισμού περιβάλλοντος. Υπάρχει παράγραφος 7 δίνονται εξηγήσει δηλαδή στα κριτικά σημεία από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην παράγραφο 22 που μιλάει για τους επισκέπτες, επιστήμονες που πληρώνονται. Τρεις ήταν το 2010 και χωρίς να έχουν πληρωθεί μάλιστα. Ούτε καν αποζημίωση δεν πήρανε, ούτε τίποτα άλλο από τον οργανισμό. Αυτό αποδεικνύει την ποιότητα δουλειάς που γίνεται στον οργανισμό αυτόν. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γίνεται πολύ καλή δουλειά, δεν ξοδεύουν λεφτά γι' αυτό. Οπότε, δεν την καταλαβαίνω την κριτική της εισηγήτριας. Τέλος πάντων, θα ολοκληρώσω σύντομα. Αυτό που είναι κρίμα είναι ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε στην ε, κριτική που γίνεται όσον αφορά για τα υψηλά, τις υψηλές μεταφορές, τα carry-overs. όντω. αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Δεν ξέρω, είναι υπερβολικά υψηλό ο προπολογισμό που παίρνουν οι οργανισμοί. Δεν θα πρέπει αυτό να το δει η Επιτροπή Προπολογισμών όμω. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο όντως μας απασχολεί και έχει να κάνει με, όλες, με όλους τους οργανισμούς. Συμφωνώ και για αυτά που είπε για τη ΣΕΠΟΛ ε, που λέει η κυρία Μακοβέη. Πριν από δύο χρόνια είχαμε σημειώσει τέτοιες επικριτικές παρατηρήσεις. Εγώ συμφωνώ η ΣΕΠΟΛ να πάει με την Ευρωπόλ, δεν βλέπω γιατί να μην πάει. Τώρα περιμένουμε το λεκτικό συνέδριο να μας συμβουλέψει γι' αυτό με μια γνωμοδότησή του. Αυτά, τίποτα άλλο, Πρόεδρε. Πρόεδρος, ο κύριος Γκάιερ. Θα είμαι πολύ σύντομος, ε, κύριε Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ και επαυξάνω με αυτά που είπαν οι κύριοι Χέρτσοκ και Γκεμπράντι. Ε, για αυτή την τόσο ε, επίμαχη έκθεση. Αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να δώσουμε στους οργανισμούς τους οποίους επικρίνουμε τρεμήτατα να αντιδράσουν στις αιτιάσει. Βέβαια δεν έχουμε πολύ χρόνο μέχρι το μεσημεριανό διάλειμμα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό ε, στους ε, συντονιστές. πώς ε, πρέπει το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης να το επανεγγράψουμε. Ε... δύο θα μιλήσουν ο Σεφμάς πρώτον που εκπροσωπεί τον έκαλο. Νομίζω ότι είναι και συντονιστή για άλλους του οργανισμούς. Και μετά η κυρία Κλέιτσε, νομίζω το προφέρω καλά, που είναι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Όσο γίνεται πιο σύντομα. Ξέρω ότι σας ζητάω κάτι δύσκολο, αλλά ε, ξεκινήσαμε με καθυστέρηση και πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα. Παρακαλώ, κυρία Μάης, έχει το λόγο. Α, ο κύριος Μάης μάλλον. Πού είναι. Α, εκεί, ναι. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητή κυρία εισηγήτρια, αγαπητά μέλη. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε ως συντονιστής του δικτύου να μπορούμε να μπορώ και εγώ να απαντήσω σε αυτό το σχέδιο για την απαλλαγή των οργανισμών. Υπάρχουν εδώ αρκετοί συνάδελφοι. Ε, γνωρίζω ότι μπορούν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις που ενδεχομένως προκύψουν. Γνωρίζω επίσης ότι και αργότερα είναι στη διάθεσή σας ε, για σχόλια ε, το οποίο ενδεχομένως θα επιθυμούσατε ε, να κάνετε. Επίσης, ε, ξέρω ότι πολλοί συναδελφοί δεν μπόρεσαν να έρθουν σήμερα εδώ, αλλά παρακολουθούν τη συνάντηση μέσα από το web streaming. Και γι' αυτό σας παρακαλώ να πούμε ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι εξετάσατε το θέμα των οργανισμών ως προκατακτική παρατήρηση θέλω να πω το Όλοι οι οργανισμοί συστήθηκαν με νομοθετική πράξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Και είναι απόλυτα υπόλογοι οι οργανισμοί στους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφέρουν υπηρεσίες στους οργανισμούς, στους πολίτες και γι' αυτό το λόγο συστήθηκαν με νομοθετική πράξη. Κατόπιν τούτου οι οργανισμοί έχουν λάβει εντολή σύστασης. Ε, βέβαια υπόκεινται σε πολύ αυστηρό έλεγχο, πολιτικό, οικονομικό και επίσης ε, η λειτουργία τους ε, ελέγχεται συστηματικά και από εσωτερικούς και από εξωτερικούς ελεγκτές. Έχοντας όλα αυτά κατά νου, οι οργανισμοί πιστεύουν ότι το ύφος του σχεδίου της έκθεσης μπορεί να τύχει παρερμηνιών και πιστεύουν επίσης ότι εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος η έμφαση να αποδοθεί περισσότερο ε, σε κινδύνους και όχι σε πραγματικά αποτελέσματα στα οποία κατέληξε το ελεγκτικό συνέδριο. Όπως ε, είπε και ο Σνάλφος από το ελεγκτικό συνέδριο, οι οργανισμοί ε, είναι ε, υπόλογοι για τα σχόλια που γίνονται ε, έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οποτεδήποτε εντοπίζονται δυσκολίες ε, στον οικονομικό ή σε άλλο διαχειριστικό τομέα οι οργανισμοί και ο κάθε μεμονωμένος οργανισμός θα κάνει ό,τι μπορεί για να επιτύχει βελτίωση. Τώρα, την άποψη που έχουν αρκετοί συνάδελφοι ότι προκύπτουν δυσκολίες αυτές ε, πράγματι σε ορισμένες περιπτώσεις ε, υπάρχουν ουσιαστικές δυσκολίες. Οι οργανισμοί είναι ανεξάρτητοι, έχουν μια οικονομική αυτοδιάθεση, γι' αυτό είναι λυπηρό το γεγονός ότι το ύφος της έκθεσης καταλήγει στο ότι οι οργανισμοί ε, λειτουργούν με μη επαγγελματικό και μη διαφανή τρόπο. Οι οργανισμοί προσβλέπουν στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και ε, ελπίζουν ότι θα δοθεί μια ρεαλιστική εικόνα για το πώς ακριβώς ε, ε, χρησιμοποιούνται τα κονδύλια που διατίθενται στους οργανισμούς. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του συντονιστικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Χημικού Οργανισμού εμείς θα παραδώσουμε στον επόμενο οργανισμό που θα είναι αρμόδιος ε, και νομίζω ότι θα υπάρχει σίγουρα κάποιος ε, συντονιστής ε, που θα, στον οποίο θα μπορούν να απευθυνθούν τα μέλη. Εδώ θα ήθελα να σταματήσω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και θα ήθελα να ζητήσω από την επόμενη συνάλφο, από τον Οργανισμό Περιβάλλοντος, να συνεχίσει. Ευχαριστούμε κυρία Γλέτς. Εσείς ε, ακούσατε και τον κύριο Κεμπραντρή να μιλάει για τη, το δικό σας οργανισμό και έχετε να πείτε εσείς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω σύντομα την, στο σχέδιο έκθεσης και να αναγνωρίσω τη σημασία της δουλειάς σας. Αυτά προσβλέποντας στη συνάντησή μου με την εισηγήτρια αύριο. Η απάντηση των υπηρεσιών έχει διανεμηθεί στα μέλη και τονίζει ότι αυτά που λέγονταν σε εννέα παραγράφους για παρατυπίες και ατασταλίες δεν έχουν τελικά αποδειχθεί από το συνέδριο. Αυτό το λέω στεναρά γιατί η φήμη των υπηρεσιών αυτών πλήτεται αλλά όποτε ακούγονται κατηγορίες χωρίς βάση αυτό πλήττει και την αξιοπιστία ολόκληρης της Ένωσης. Ελπίζω με να λυθεί αυτό και το συνέδριο να το αναγνωρίσει. Το σοβαρότερο όμως θέμα που θέλω να θίξω είναι το ότι θεωρείται ότι μερικές υπηρεσίες έχουν αναλάβει και δράσεις άσχετες με το θέμα τους λέγεται ότι υπάρχει έλλειψη ανταπόκρισης μεταξύ δράσης των υπηρεσιών και στόχου τους. Αυτό δείχνει μεγάλη έλλειψη κατανόησης και γνώσης για τη δουλειά μας. Αλλά και μέλη της Επιτροπής της Κομισιόν, δηλαδή και η εισηγήτρια δεν το δέχονται αυτό θεωρούν ότι η χρήση των επιχορηγήσεων από την Ένωση είναι κάτι που το έχει προβλέψει ο ίδιος ο νομοθέτης και δεν αποτελεί παρατυπία. Για τα τελευταία πέντε χρόνια ακόμη και εκπρόσωποι της βιομηχανίας έχουν επενέσει τη λειτουργία των υπηρεσιών για την πληροφόρηση των ε, εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Σε άλλα μέρη του κόσμου οι υπηρεσίες σαν τη δική μας του περιβάλλοντος δηλαδή επίσης την χάνουν επικρίσεων και επιθέσεων από όσου έχουν συμφέροντα. Γι' αυτό θα ήταν ζωτικό για την Επιτροπή σας να καταλάβει ποια είναι η βάση αυτών των επικρίσεων. Η Ευρώπη ωφελείται πολύ από την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουν οι νομοθέτες στις πληροφορίες που διαθέτουν και το να την καταστρέφουν αυτή την εμπιστοσύνη με βάση λανθασμένες πληροφορίες είναι κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Παραδείγματος χάρη, οι διαπραγματεύσεις για το περιβάλλον και οι εκθέσεις για τις εκπομπές διοξιδίων είναι πράγματα που αφορούν και ενδιαφέρουν ολόκληρο τον κόσμο και συνδέονται με τη στρατηγική του 2020 αν δεν τροπολογηθεί η έκθεση αυτή τότε θα βλαφτεί μόνιμα το κύρος και η αξιοπιστία των υπηρεσιών ακριβώς τη στιγμή που προσπαθούν να γίνουν ηγέτες στον κόσμο για τις πρωτοβουλίες όπως τη μείωση των εκπομπών. Θα ήθελα με τις τροπολογίες τους να εξισορροπήσουν την έκθεση οι βουλευτές για να ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα. Τελειώνω εδώ ελπίζοντας να μην καταστραφεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι υπάρχουν εδώ και άλλοι εκπρόσωποι από διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που θα θέλαν να πάρουν το λόγο. Αλλά βλέπετε είμαι αντιμέτωπος με το χρόνο. Είχαμε αντιδράσει όμω, γραπτέ από διάφορου Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Θα του βάλουμε όλε αυτέ τι παρατηρήσει μαζί, θα τι συζητήσουμε στου συντονιστέ, με του συζητητέ και τους σκιώδες συζητητέ. Ό,τι υπάρχει γραπτά δηλαδή, τα λέει όλα. Οπότε δεν θα αλλάξει τίποτα, σα δώσω τώρα το λόγο για ένα-δύο λεπτά. Η συζήτηση θα γίνει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Η κυρία Μακοβέη έτσι κι αλλιώ ηγείται του θέματο αυτού είναι σε επαφή με τους ε, εισηγητές, με τους σκιώδους εισηγητές. Οπότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Μακοβέη, το λόγο για να κλείσει αυτό το θέμα, να μπορέσει να απαντήσει στις διάφορες ερωτήσεις που της τέθηκαν. Και ζητάω από τους διερμηνείς πέντε λεφτά παρακαλώ παραπάνω, ώστε να μπορέσει η κυρία Μακοβέη να ολοκληρώσει. Yes, thank you. Um... Μάλιστα. για τη συνεργασία με τους Κιώδης. Πρόκειται για πρόοδο σε σύγκριση με πέρυσι όπου δεν είχαμε καμία τέτοια συνεργασία. Έχουμε ήδη συναντηθεί και είχαν πρόσβαση και στο λεγόμενο εμπιστευτικό έγγραφο. Λοιπόν, από την πλευρά μου θα συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί τους. Και αναμένω βέβαια τις τροπολογίες τους. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω το θέμα της διαμάχης συμφερόντων με υπηρεσίες που συνδέονται με βιομηχανίες. Χρειάζονται, λέει, εμπειρογνώμονες και δεν μπορούν να τους βρουν παρά μόνο στη βιομηχανία. Εδώ όμως θα ήθελα να πω ότι εδώ είναι και ο κίνδυνος. Πρέπει να το προσέξουν αυτό. Θα μπορούσαν, αν κάποιος έρχεται από την εταιρεία Α στην υπηρεσία να μην που πιστοποιεί φάρμακα να μην του βάλουν την ίδια δουλειά που είχε και στη βιομηχανία του για να αποφευχθούν έτσι οι διαμάχες. Τελεία. Υπήρξε κάποιο ανάλογο πρόβλημα με την ασφάλεια της αεροπλοείας. Για την υπηρεσία περιβάλλοντος θα συναντήσω αύριο τον διευθυντή. Προσπάθησα και στο παρελθόν αλλά δεν το καταφέραμε. Αλλά θα ήθελα να σχολιάσω Πρόκειται για την άποψή μου και ο κάθε συνάδελφος έχει την ελευθερία να καταθέσει τροπολογίες και οι υπηρεσίες να την επικρίνουν, αλλά αφού μιλάμε για την υπηρεσία περιβάλλοντος, δυστυχώς δεν ελέγχει τα στοιχεία που δίνουν τα κράτη-μέλη, δεν έχει ρυθμιστικές δικαιοδοσίες και βασικά απλώς γράφει εκθέσεις. Βεβαίως και άλλα σώματα γράφουν εκθέσεις και ίσως θα έπρεπε να δούμε με αυτό το κριτήριο την υπηρεσία αυτή και τις επόλοιπε. Η υπηρεσία για την ισότητα των φύλων ήταν η τελευταία που δημιουργήθηκε. Δεν θέλω να τη σχολιάσω αυτήν συγκεκριμένα, αλλά Έχουμε ήδη μια υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν μπορεί, και αυτή, να, δεν μπορεί αυτή να καλύψει και το θέμα της ισότητας των φίλων. Γιατί χρειαζόμαστε χωριστή υπηρεσία και προπολογισμό. Υπάρχουν λοιπόν θέματα που πρέπει να εξετάσουμε για να δούμε πώς θα πανώνται τα χρήματα. Επίσης, πολύ σύντομα, η αξιοπιστία των υπηρεσιών, όπως είπε η υπηρεσία περιβάλλοντος, η αξιοπιστία τους δεν ταυτίζεται με την αξιοπιστία της Ένωσης. Η αξιοπιστία της Ένωσης σημαίνει και σωστή διαχείριση και εξοικονομήσεις. Εδώ ζητούμε από τον κόσμο να μειώσει τα έξοδά του, ε, το ίδιο πρέπει να ζητήσουμε και από τις υπηρεσίες όχι συνεχώς αύξηση των δαπανών τους ή μέτρα λιτότητας μόνο για τον κόσμο. Κάποτε ίσως υπήρχαν λεφτά και λέγαμε ας δημιουργήσουμε την α και τη β υπηρεσία αλλά τώρα πρέπει να σκεφτούμε αν τις χρειαζόμαστε όλες ή όχι και με τον ίδιο προϋπολογισμό. Ευχαριστούμε. Τελείωσε εδώ η συνεδρίασή μας για σήμερα το πρωί και ευχαριστώ πολύ τους διερμηνείς που μας έδωσαν 10 λεφτά και παραπάνω, ειλικρινά. Ε, συνεχίζουμε στις 3, αλλά όχι σε αυτή την αίθουσα. Προσοχή, έτσι, πάρτε τα χαρτιά μαζί σας. Δεν συνεχίζουμε σε αυτή την αίθουσα, αλλά στην αίθουσα 4Β001, στο Πολ Ανρί Σπακ. Θα τα ξαναπούμε τότε.